Το 2011, όπως προβλέπετο, δημοσιεύτηκε η έκθεση. Η Κομισιόν είχε κάποια δυσκολία να συλλέξει συμβολές και συνεισφορές για αυτήν. Το αίτημα εστάλει στα κράτη-μέλη, στις υπηρεσίες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2011 ε, και αν και η προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, ε, η Κομισιόν έλαβε μόνο ένα τμήμα των ε, συνεισφορών. Το Σεπτέμβριο είχε λάβει 25 συνεισφορές για να γίνει έκθεση. Παρά τις καθυστερήσεις, η Κομισιόν κατάφερε να δημοσιεύσει έγκαιρα την έκθεση αυτή δεν υπάρχει συγκεκριμένος μορφότυπος. Η Κομισιόν ε, είχε ένα ε, έγγραφο εργασία ε, σχετικά με την υποβολή της έκθεσης. Σε αντίθεση με το 2009 η έκθεση δεν, είχε, δεν ήταν ως συνημένη, σε, κάποια ανακοίνωση. Ε, διότι ε, υπήρχαν κάποιες, ε, η ατζέντα για την αλλαγή η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για την συνοχή της πολιτικής. Δεν υπάρχουν προτάσεις για αλλαγή πολιτικής στην ατζέντα και γι' αυτό είναι απόλυτα ίση η μορφή του, της υπηρεσιακής αυτής έκθεσης, του υπηρεσιακού εγγράφου. θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή ε, μετά την έκθεση αυτή του 2009. Η κυρία Σνίμπερ Γιάστραμ θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, θα ήθελα να ξέρω αν αληθεύει ότι το θέμα PCD στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ε, θα παραμείνει ή θα, αν θα, παραμείνει στο ίδιο τμήμα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης ή αν θα πάει σε άλλο. Η ομάδα αυτή και το PCD Development θα είναι στην ε, Γενική Διεύθυνση Α Γενικής Πολιτικής. Ε, μεταφέρεται από την ε, μονάδα Α3 στην μονάδα Α1. Η κυρία Κέλλερ δεν είναι εδώ, δεν μπορούμε λοιπόν να τη ρωτήσουμε, αλλά στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην οποία την Προεδρία έχει ο κύριος Ντέβα, ακούσαμε μια ερώτηση για την οποία σας ζητήσαμε να μας δώσετε μια απάντηση σήμερα. Είναι οι σχέσεις ε, μεταξύ ΕΣΕΡ και ΝΤΕΦΚΟ, είναι η ερώτηση της 8ης ε, Δεκεμβρίου και θα ήθελα να μου πείτε αν για το θέμα αυτό της SEA ή e έχετε κάποια απάντηση να μας δώσετε. Ε, Η συμφωνία για την εργασία υπεγράφει στις 13 Ιανουαρίου μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και του ε, επικεφαλής ε, ε, στο ΙΕΣ για τον τρόπο εφαρμογής της συνεργασίας μεταξύ της υπηρεσίας και των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής. Ε, συνθήκες εργασίας ε, για τις αντιπροσωπείες, για συνεργασία σε περίπτωση κρίσης ε, και σχέσεις μεταξύ γραφείων ΕΚΟ και των αντιπροσωπιών, την επικοινωνία στα ΜΜΕ και τις ενημερώσεις. Προβλέπεται ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων είναι αποκλειστική ευθύνη της Κομισιόν και το ΙΕΣ e παίζει μεγάλο ρόλο για τον προγραμματισμό των μεγάλων μέσων και αναφέρεται λεπτομερώς πώς αλληλεπιδρούν οι Κομισιόν και η ΙΕΣ. E Με περισσότερες λεπτομέρειες η ΙΕΣ e παίζει ε, ηθήνοντα ρόλο στον προγραμματισμό EDF και DCI υπό την ευθύνη του Επιτρόπου Ανάπτυξης και τα διάφορα βήματα στην προγραμματική διαδικασία, τη διαδικασία προγραμματισμού είναι ότι το ESS, η συμφωνία με την Κομισιόν, κάνει, ε, υποβάλλει προγράμματα στις αντιπροσωπείες. Ε, μετά οι αντιπροσωπείες επιτόπου αρχίζουν διαβουλεύσεις με τη χώρα εταίρο και στέλνουν τέλος τις προτάσεις τους ε, για τα έγγραφα στρατηγικής στο EuroPaid και στο ES. Ε, οι συναντήσεις των ομάδων σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή ΙΕΣ και Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών και άλλων ενδιαφερομένων υπηρεσιών αξιολογούν τις προτάσεις και μετά ε, η ομάδα υποστήριξης, στήριξης της ποιότητας ε, διυπηρεσιακά κάνει το ίδιο υπό τις ΙΕΣ και EuroPaid. Οι διαβουλεύσεις διυπηρεσιακά για να οριστικοποιηθεί η πρόταση της Κομισιόν αρχίζει από την ΕΕ σε, συνεργασία, σε συμφωνία με την ε, EuroPaid. Μετά η πρόταση πηγαίνει στην αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου, όπου η EuroPaid προεδρεύει και παρέχει η γραμματεία και η ΕΕΣ παρουσιάζει τις προτάσεις και απαντά σε ερωτήσεις των κρατών μελών. Η και η από κοινού απαντούν ε, στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ε, για το DCI. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Τέλος, το ΙΕΣ είναι υπεύθυνο για την υποβολή της γραπτής, την έναρξη της γραπτής διαδικασίας για την τελική έγκριση από την Κομισιόν, οπότε οι ε, ρυθμίσεις εργασίας μπαίνουν σε αρκετές λεπτομέρειες, ούτως ώστε να δώσουν σάρκα και ωστά στην απόφαση του Ιουλίου του 2010 ότι τα έγγραφα αυτά από κοινού προετοιμάζονται από την ΙΕΣ και τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Ίσως ό,τι αφορά τα θεματικά προγράμματα, η Europe Aid, παίζει πρωτεύοντα ρόλο για τα, τον προγραμματισμό και η ΕΣ είναι συμβουλευτική στις, στα βήματα των διαδικασιών. Για την εφαρμογή, για τα μέσα, τα προγράμματα, τα ετήσια προετοιμάζονται από την ε, Europay που ε, και γίνονται υπηρεσιακές ε, διαβουλεύσει, υποβάλλεται στη διαδικασία τη επιτροπολογία σχέδιο και αρχίζει έτσι η διαδικασία έγκρισης από το κολέγιο. Η εφαρμογή επίση είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα της γενική διεύθυνση Europay, ενώ η ΕΣ συμβάλλει μέσα από του επικεφαλεί αντιπροσωπείων που δρούν επιτόπου ω διατάκτες. Να ρωτήσω και εγώ, εάν ε, οι δύο οργανισμοί δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους, οι αποφάσεις για τα ετήσια προγράμματα και τον προγραμματισμό γενικώ λαμβάνονται σε επίπεδο συλλογικού σώματος, κολεγίου. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Όχι. Κύριε Γκέρενς, η ερώτησή μου συνδέεται άμεσα με αυτό που είπατε. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το συντονισμό. Ποιος φροντίζει να συντονίζονται μεταξύ τους πολιτικές των κρατών μελών. Τα θέματα ανάπτυξης είναι η Europaid. Είναι ένας από τους ρόλους που έχει αναλάβει η υπηρεσία Α1, Α1, όπως το είπαμε. Είναι ένας από τους ρόλους της Επιτροπής μας στην αναπτυξιακή πολιτική. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Αν και έχω την αίσθηση ότι δεν λάβατε απάντηση, κύριε Γκέρενς. Δεν φαίνεστε ικανοποιημένο. Νομίζω ότι το ερώτημα σωστά έτεθη και είναι και εύστοχο αλλά θα παραμένουμε διαρκώ ανικανοποιητοί εφόσον δεν αλλάξει το πλαίσιο και δεν έχουμε μια συζήτηση και κλεισμένων των θυρών, ώστε να μπορεί ο καθένα να πει αυτό που πραγματικά σκέφτεται. Έτσι δημοσίω δεν έχει πολύ νόημα, διότι σε κάθε περίπτωση ο καθένας λαμβάνει κάποιες ρητορικές ε, μέρημνες όταν τοποθετείται και όλοι μένουν ικανοποιητές. Στην επόμενη λοιπόν συνάντηση των συντονιστών Και επειδή μιλάμε για την αποτελεσματικότητα, τη θεσμική αποτελεσματικότητα τη ευρωπαϊκή προσέγγιση στο σχετικό θέμα, καλό θα ήταν να τον δούμε. Πρόεδρο, μάλιστα, θα το συμπεριλάβουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, σύντομα κιόλα, μια συνεδρίαση κυκλισμένων των θυρών με του συντονιστέ. Σημειώθηκε. Θα γίνει. Πολύ ωραία. Δεν φαντάζομαι ότι αγνοεί κανεί ότι η έκθεση που ετοιμάστηκε για την συνοχή των αντιξιακών πολιτικών για την τελευταία διετία λαμβάνει στοιχεία από βάσει δεδομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, τη κοινωνία των πολιτών και το Ευρωκοινοβούλιο. Επίση, υπάρχει το άρθρο 208 τη Συνθήκη τη Λισαβόνα, που σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ δεν επηρεάζουν αρνητικά τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Και αναθέτει στην Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων να ε, δημοσιεύσουν έκθεση για το ίδιο θέμα με σκοπό να αποτιμήσουν τι διάφορε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την έκθεση του 2009, η νέα έκθεση αφορά την επισκεπτική ασφάλεια, του φυσικού πόρου, την ε, ασφάλεια των πολιτών και την μετανάστευση. Πάντοτε σε συνάρτηση με τι αναπτυξιακέ πολιτικέ. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Concord, με την ε, παρουσία τη μόνιμη συζητριά μα για το θέμα, τη κυρία Σνίμπερ Γιάστραμ, είναι ένα πρώτο στάδιο για την ετοιμασία έκθεση πρωτοβουλία με σκοπό να ετοιμαστούν κάποιε συστάσει για αυτό το τόσο σημαντικό τομέα. Να δώσω λοιπόν το λόγο αρχικά στον εκπρόσωπο τη ε, Concord και στην εκπρόσωπο τη ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ για τι ε, παρουσιάσει του και μετά θα έχουμε συζήτηση με του συναδέλφου. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο τη Concord, τον κύριο Γιάννησεν, για 10 λεπτά. Well, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. I don't know if you're able to see my PowerPoint presentation. Well, let me start off. Ε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή ΔΕΒΕ. Πριν αρχίσω να παρουσιάζω την έκθεση, θέλω να, καλωσορίσω, να χαιρετήσω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβάλει έκθεση και με μόνιμο εισηγητή φέτος για την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Ως Concord προσβλέπουμε στην έκθεση αυτή και τώρα με την Προεδρία της Δανίας η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής είναι πολύ σημαντικό πράγμα και είναι κομμάτι της, του επίσημου προγράμματος Δανικής Προεδρίας και είναι σημαντικό ε, σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών. Όπως είπε και η Πρόεδρος ε, πριν, η έκθεση Well, continue. Yeah. The foundation of... Η βάση της έκθεσης είναι οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, άρθρο 208, σχετικά με την ε, συνοχή των πολιτικών για τις αναπτυσσόμενες χώρες και είναι πάντα σημαντικό να Μπορούν να χαμηλώσουν τα φώτα. Ευχαριστώ. Συνεχίζω λοιπόν, εδώ είναι το άρθρο 208 σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους που ενδεχομένως επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι ο απότερος στόχος της χρήσης αυτών των πολιτικών είναι η εξάλληψη της φτώχειας. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αντίκτυπος θετικός ή αρνητικός, αυτό βλέπουμε, ε, σε σχέση με την επίτευξη του στόχου εξάλληψης της φτώχειας. Κάποια ψηφίσματα κοινοβουλίων ήδη αναφέρουν τις αρχές που διέπουν τα διάφορα θέματα και τις νομοθετικές διαδικασίες. Ήδη το καλοκαίρι φέτος είχαμε το ψήφισμα ε, για την ΚΑΠΑ, για την επισητιστική ασφάλεια και για τις πρώτες ύλες ε, ειδικά ε, αναφερόμενο στα θέματα των αναπτυξιακών στόχων στα πλαίσια της εξέλιξης και προόδου στον δημοκρατικό έλεγχο που πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή. Η δική μας η προσέγγιση στην έκθεση της Concord ε, στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της θα έχουν συνοχή με την εξωτερική δράση και αντίκτυπο των πολιτικών της σε συνδυασμό με τα βασικά της, ε, ε τις βασικές της αρχές, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, που επίσης υπάρχουν στη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτό το βλέπουμε ως μια έξω υποχρέωση που ενδυναμώνει δικαιώματα ε, των πολιτών πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Δεν βλέπουμε το στόχο της εξάλληψης της φτώχειας, ε, δεν βλέπουμε πόσο στόχος εξάλληψης της φτώχειας μπορεί να εξαλειφθεί χωρίς να ενδυναμωθούν τα δικαιώματα των πολιτών εκτός Ευρώπης. Τώρα, το, η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής ε, τι ρόλο παίζει ως ε, ε, εργαλείο. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι τώρα η διασύνδεση μεταξύ των περιοχών του κόσμου αυξάνεται και οι εξελίξεις εκτός Ευρώπης και η ανάπτυξη εκτός Ευρώπης εξυπηρετεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης. Και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να ενσωματωθεί στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι οι πολιτικές της Ένωσης θα είναι διαφανέστερες και θα υπάρχει μια γενικότερη ε, συνολική νομιμοποίηση. Είναι επίσης αυτός ένας τρόπος ε, για να είναι πιο συμμετοχική η διαμόρφωση της πολιτικής και η διακυβέρνηση θα ανταποκρίνεται στους εμπλεκόμενους εκτός Ευρώπης και θα λαμβάνει υπόψη και τους περιθωριοποιημένους στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ε, είναι σημαντικό να υπάρχει λογοδοσία προς τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρησιμοποιούνται με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο και να μην καταστρέφουμε με το ένα χέρι αυτό που φτιάξαμε με το άλλο. Η μέθοδος που ακολουθεί η έκθεση, όπως είπα, στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα για την ανάπτυξη. Τι κάνουμε εδώ, Έχουμε τέσσερα θεματικά κεφάλαια στην έκθεση που εστιάζουν στα διάφορα δικαιώματα όπως δείχνει το παράδειγμα εδώ, το δικαίωμα στα τρόφιμα, ένα δικαίωμα που ε, κατοχυρώνεται σε διεθνείς συμβάσεις αλλά ε, γίνεται λειτουργικό και στα 175 κράτη του κόσμου και τη, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, πώς μπορεί να εφαρμοστεί το δικαίωμα αυτό για τους φτωχούς εκτός Ευρώπης. Αρχίζουμε να χαρτογραφούμε. Ποιες είναι οι πολιτικές που επηρεάζουν το δικαίωμα αυτό και την εφαρμογή του. Η εμπορική πολιτική, η πολιτική για το κλίμα, η κοινή αγροτική πολιτική, για παράδειγμα, που έχουν με διάφορους τρόπους αντίκτυπο στη δυνατότητα ε, ε, πραγματοποίησης του δικαιώματος. Και αυτή η προσέγγιση, η δομή, κάθε κεφάλαιο που ε, έχουμε για τις διάφορες πολιτικές και αξιολογείται κάθε φορά ο αντίκτυπος των πολιτικών μας. Τώρα, δύο παραδείγματα. Μία μελέτη περιπτώσεων καταρχήν, που ε, έχουμε περίπου 12 περιπτωσιολογικές μελέτες στην έκθεση, μπορείτε να τις δείτε λεπτομερώς, αλλά για να πάρουμε ένα παράδειγμα. Μία μελέτη για το δικαίωμα στα τρόφιμα, για εξαγωγές γάλατος σε σκόνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα έχουμε κρίση πείνας ε, πάρα πολλοί πηγαίνουν στο κρεβάτι πεινασμένοι και πάνω από ένα τρίτο των χωρών ε, σήμερα σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ανασφάλεια στα τρόφιμα και ξέρουμε ότι η μόνη διατηρήσιμη λύση μακροπρόθεσμα για να λυθεί το πρόβλημα είναι να επιτρέψουμε την ανάπτυξη τη γεωργική τοπικά, εκεί στις χώρες που ζουν οι φτωχοί και οι πεινασμένοι. Το γάλα και τα γαλακτοκομικά θεωρούνται από και η παραγωγή τους είναι από τις πιο σημαντικές απασχολήσεις. Έχουμε 750 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από τα, τον τομέα των γαλακτοκομικών, την ενασχόληση εκεί. Επίσης έχει πολλές θεμητές πολιτικές η Ένωση για να ε, προωθήσουν ε, τον τομέα αυτό στην Ευρώπη, αλλά καμιά φορά μπορεί να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αντέδρασε στην κρίση της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πανισάγοντας εξαγωγικές επιστροφές ε, και έγιναν αγορές αξίας 6 εκατομμυρίων για αγορά φρέσκου γάλατος για να γίνει σκόνη. Στην υποσαχάρια Αφρική οι εξαγωγές ε, από την Ένωση αυξήθηκαν ε, κατά 62% και αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά ε, τους ντόπιου παραγωγούς αυτές οι μεγάλες εισαγωγές της χώρες αυτές και να αλλάξουν τα δεδομένα. Στο Καμερούν, για παράδειγμα, είδαμε ότι οι αγρότες που επί 10 χρόνια ε, είχαν εκρεώσει τη θέση τους ε, στην ε, αλυσίδα του εμπορίου, παραγωνίστηκαν λόγω των εξαγωγών από την Ένωση. Και στο Μπαγκλαντές συνέβη κάτι παρόμοιο και σε άλλες χώρες βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς οι πολιτικές της Ένωσης επηρέασαν αρνητικά την δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το δικαίωμα αυτό στα ε, τρόφιμα και στην επισητιστική ασφάλεια στην, ε, εκτός Ευρώπης. Τώρα, ε, φοροδιαφυγή... Η Γκλέγκο, μια μεγάλη εξορρυκτική βιομηχανία, καλύπτει στη Ζάμπια τις περισσότερες εξορυκτικές δραστηριότητες και μια έκθεση που διέρευσε έδειξε ότι για χρόνια ε, τεχνιέντος έδιωχναν τα κέρδη από τη Ζάμπια υπονομεύοντας έτσι τη φορολογική βάση της χώρας αυτής. Αυτό είναι ένα παράδειγμα επίσης παγκοσμίου προβλήματος αφού υπολογίζεται ότι ε, η οχταπλάσια ανάπτυξη από αυτή που ε, ε, ε, από αυτή που πραγματοποιούμε φεύγει έξω από τη χώρα αφού πολλές πολυεθνικές βγάζουν σε φορολογικούς και πάνε σε φορολογικούς παραδείσους τα κέρδη τους. Αυτό έχει να κάνει με το λογιστικό σύστημα της Ένωσης όπως έχει τώρα η νομοθεσία μας. Οι εταιρείε δεν χρειάζεται να υποβάλουν έκθεση σε κάθε χώρα αλλά υποβάλλουν οικονομική έκθεση συνολικά. Άρα δεν βλέπετε πόσο κερδίζουν και πόσους φόρους πλήρωσαν στις χώρες όπου λειτουργούν. Αυτό είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία και φαίνεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα αλλάξει τώρα προς το καλύτερο. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα όμως που ε, ε, δείχνει ότι οι εσωτερικοί κανόνες της Ένωσης επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη τον κόσμο που ζει στι αναπτυσσόμενες χώρες. Κάποια συνολικά ευρήματα τη έκθεσης τώρα δείχνουν όπως δείχνουν και αυτές οι περιπτώσεις και άλλες όμως, ότι πολλές νέες ευρωπαϊκές πολιτικές δεν συνάδουν με τους αναπτυξιακούς στόχους. Αλλά Υπάρχει ε, περιθώριο βελτίωσης στους υφιστάμενους μηχανισμούς για το, από το 2009 και μετά, για παράδειγμα, οι κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης ε, για τις μελέτες επιπτώσεων δείχνουν ότι κάθε μελέτη επιπτώσεων θα πρέπει να δείχνει αν θα υπάρξει αντίκτυπος στην ανάπτυξη και εξωτερικός αντίκτυπος σε νέα προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε κάνει 164 μελέτες επιπτώσεων από το 2009 77 από αυτές είχαν σχέση ενδεχομένως για τις με τις αναπτυσσόμενες, αλλά ε, λίγες αναφέρουν την ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα παράδειγμα κακοδιοίκησης ε, και σε σχέση με τους στόχους των κατευθυντηρίων. Ε, τώρα, για τους μηχανισμούς προσφυγών, εδώ ε, πιέζουμε από το 2009, τονίζοντας ότι χρειάζονται κάποιοι μηχανισμοί ώστε όσοι έχουν πληγεί στις αναπτυσσόμενες χώρες από τις ε, πολιτικές της Ένωσης να μπορούν να προσφεύγουν κάπου με την υπόθεσή τους και σε τελευταία ανάλυση όλα αυτά και οι φυστάμενοι μηχανισμοί και οι διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής στην Ένωση είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και εδώ ίσως ε, παρατηρούμε μια έλλειψη πολιτικής βούλησης. Δεν ξέρω πόσο χρόνος μου μένει ακόμη. Ε, ε, το τελευταίο που θέλω να θίξω είναι πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει, όπως είπα και στην αρχή. Τώρα στη... περιμένουμε την επόμενη έκθεση και ελπίζουμε ότι δεν θα είναι τόσο περιγραφική αν θέλετε όσο η έκθεση της Κομισιόν. Βέβαια ακούσαμε ότι υπάρχουν λόγοι για το, τη μορφή της παρούσας έκθεσης, αλλά ελπίζουμε ότι η νέα έκθεση από τον καινούριο οριστέντα εισηγητή θα είναι πιο φιλόδοξη. Ελπίζω επίσης ότι το Ευρωπαϊ... Ε, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ιδιαίτερη ευθύνη και ευκαιρία γιατί είναι συνομοθέτης. Και αυτό σημαίνει ότι σε σχέση με την νομοθεσία που διέπει την ΚΑΠ ή την νομοθεσία για το δημοσιονομικό, του δημοσιονομικό κανονισμό, υπάρχει δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει σε ε, νομοθεσίες που θα έχουν μεγαλύτερη συνοχή με τους αναπτυξιακούς στόχους. Έχετε τη δυνατότητα, κυρίως η Επιτροπή σας, να διοργανώσει ε, ακροάσεις για να βελτιωθεί ο διάλογος και να δημιουργηθεί κατανόηση πέρα από την αναπτυξιακή φούσκα επίσης και ε, εσείς είστε δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί, οπότε η πολιτική σας υποστήριξη είναι προφανώς κέρια σημασίας. Τέλος, πολύ σύντομα να χαρτογραφήσω τρεις κύριες διαδικασίες ε, που θεωρούμε ότι εκεί εμπλέκεται το Κοινοβούλιο φέτος. Ε, καταρχήν έχουμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και παρά το γεγονός ότι το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφώς αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει αναφορά στο PCD, στην ε, νομοθεσία για την ΚΑΠ, δεν υπάρχει αναφορά στην ε, νομοθεσία, μπορείτε να το αλλάξετε αυτό και ελπίζουμε να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή σας, θα ήταν πολύ καλό. Υπάρχει επίσης η ατζέντα για την αλλαγή, για την νέα αναπτυξιακή στρατηγική που πιστεύω ότι πολύ στερνά αντιμετωπίζει το θέμα PCD και η αντίδραση του Κοινοβουλίου σε αυτή τη στρατηγική είναι πολύ σημαντική και τέλος η οδηγία για τη διαφάνεια που επίσης συζητείται τώρα. Και αν διαμορφωθεί σωστά και εκείνη θα μπορέσει να ε, καταπολεμήσει το πρόβλημα της ε, ε, παράνομης φυγής κεφαλαίων από τις ανεψόμενες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές, αν έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε. Ο κύριος Γκέρινς είναι ο πρώτος. Δεν ξέρω αν η συγγήτρια θέλει να πάρει πρώτα το λόγο. Κυρία Κέλλερ, θέλετε να μιλήσετε. Äh, ευχαριστώ πολύ αξιότιμοι εκπρόσωποι της Κομισιόν, συνεργάτες της Concord. Ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ε, η PCD, η συνοχή δηλαδή της αναπτυξιακής πολιτικής, είναι από τα σημαντικότερα θέματα που διαπραγματευόμαστε τώρα και μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι θα αποτελέσει από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μας. Ε, Σήμερα δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γι' αυτό θα περιοριστώ σε κάποιες βασικές παρατηρήσεις μόνο. Ο στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας σε τελευταία ανάλυση είναι να γίνει περιττή. Η PCD αντίθετα θα παραμείνει μια πρόκληση στο βαθμό που η πολιτική μας έχει εξωτερική επίδραση. Και η PCD είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα πράγμα που άλλωστε ισχύει σε όλα τα προγράμματα εξυγχρονισμού mainstream, τα κύρια προγράμματα. Ε, χρειάζονται και επαρκείς πόροι. Μέχρι τώρα ήταν περιορισμένη για το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων ε, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την πραγματογνωμοσύνη τους και τη βοήθειά τους. Παρά τα προβλήματα είμαι πεπισμένη ότι όλο και σημαντικότερη θα είναι η PCD στο μέλλον. Γνωρίζετε ότι ζούμε σε εποχές ε, πολιτικών ανακατατάξεων. Αυτό επηρεάζει και την PCD. Η PCD είναι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Και γίνεται αναγκαιότητα η συνοχή αυτή. Γιατί, διότι καταρχήν με μεγάλη υπευθυνότητα πρέπει να χειριζόμεθα τα χρήματα των φορολογουμένων, γιατί αλλιώς πώς θα πείσουμε τους πολίτες που ε, καλούνται να, ε, σε λιτότητα μέσα στην κρίση να ε, δώσουν περισσότερους φόρους. Οι πολίτες είναι φυσικό να ενδιαφέρονται ε, για τα θέματα αυτά ε, και να αναρωτιούνται γιατί θα πρέπει να ε, πληρώνουν και για τις ζημίες που επιφέρουν οι πολιτικές για τις οποίες καλείται να καταβάλει περισσότερα. Δεν επιτρέπεται να συνεχίζουμε πολιτικές που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη στην κάθε χώρα και έτσι συμβάλλοντας στην ε, ε, μετανάστευση. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές ε, συγκρούσεις συμφερόντων. Αυτές λύνονται όταν έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική στην πολιτική μας. Ε, μόνο με συνεκτική πολιτική θα έχουμε βιώσιμες εταιρικέ σχέσεις, διατηρήσιμες με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά δεύτερο λόγο, η αναπτυξιακή συνεργασία με σαποσυνοχή πολιτικών δεν θα είναι μόνο μια πολιτική αποκατάστασης ζημιών. Μόνο μέσα, από πολιτική, μέσα συνοχής θα δοθεί στις χώρες αυτές η ευκαιρία για αυτόνομη ανάπτυξη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς και οι αναπτυσσόμενες χώρες αλληλοεξαρτώμεθα και θα πρέπει να, καταλα... να δούμε πώς ε, θα συμβάλλουμε στο μέλλον που θα επηρεάζει και τους δύο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια βιώσιμη πολιτική. Οι πολιτικές ανακατατάξεις όμως επηρεάζουν και σε ένα δεύτερο επίπεδο τη συνοχή πολιτικών. Στην πολιτική, όπως και στην πολιτική περιβάλλοντος και έτσι και εδώ η επίγνωση των προβλημάτων δεν επαρκεί για να αλλάξει ε, μια παγιωμένη πράξη. Μετά την έκθεση «Όρια της ανάπτυξης» ε, ε, και στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις. Το 2010 ήταν το έτος ε, όπου ε, σημειώθηκε η υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το PCD. Τα προβλήματα είναι γνωστά, κυρίως μεταξύ ημών, αλλά πολύ συχνά λείπει η πολιτική βούληση για αλλαγή αγκιστρωνόμεθα και αυτό το βλέπω εγώ ως νέα ευρωβουλευτής με τρόπο ιδιαίτερα συνταρακτικό, αγκιστρωνόμεθα σε παλιές βεβαιότητες, ε, παλιά συστήματα, το βλέπουμε ίσως όταν συζητάμε με τους πολιτικούς υπεύθυνους ε, για το εμπόριο, για τη γεωργία και σε πολλούς άλλους τομείς, ε, αλλά αυτή η παγιωμένη ε, αντίληψη είναι λάθος. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία ε, να αλλάξουν οι παλιές βεβαιότητες, οι πρακτικές οι παλιές να αμφισβητηθούν και να υπάρξει ένα καινούριο καθαρό, ε, μια καθαρή προσέγγιση στα προβλήματα. Ε, σίγουρα και στο μέλλον θα έχουμε διαπληκτισμούς και με άλλες επιτροπές και με την Κομισιόν. Καλό όμως είναι αυτό, γιατί κάθε όργανο θα πρέπει την πολιτική για την οποία είναι υπεύθυνο να την ε, τάσει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, τα επιχειρήματά μας μεσοπρόθεσμα είμαι βεβαία ότι θα εισακουστούν περισσότερο. Είναι καλό δείγμα η επιτυχία στην πολιτική αλίας και αν δω την πατρίδα μου και το Βερολίνο, βλέπω ε, γεωργούς να κατεβαίνουν στο δρόμο και αυτό νομίζω ότι αποτελεί ε, μια ακόμα συμβολή στη συζήτηση. Η PCD είναι μια απόλυτη αναγκαιότητα πλέον και αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό θα μας ξεπεράσει η ιστορία. Ε, δεν μπορούμε... Α, ε, είμαι από το Αμβούργο, ε, γι' αυτό θα ήθελα να ε, αναφερθώ στη, στη θάλασσα και τους ανέμους της. Ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ούριο άνεμο στα πανιά μας. Τέλος, να ευχαριστήσω για την έκθεση της Επιτροπής και την έκθεση της Concord. Για τις δύο εκθέσεις θα ήθελα να πω ότι δυστυχώ είναι υπηρεσιακό το έγγραφο τη Κομισιόν, το ανέφερα και στην ερώτηση. Τώρα για την έκθεση της Concord, νομίζω ότι οι προτάσει σα είναι πολύ καλέ. Αναφέρει στον Παρόζο, θεματοφύλακα των συνθήκων, την Κομισιόν, θέματα του ε, διαμεσολαβητή. Ε, ε, ίσως θα πρέπει ορισμένα θέματα να λυθούν από τον πρόεδρο ή τους αντιπροέδρους μας. Σημαντική είναι η μελέτη περιπτώσεων και το θέμα των πρώτων υλών αναφέρεστε σε θέματα φορολογίας, ε, για τη διαφάνεια επίσης ε, τα κριτήρια για την πιστοδότηση θα πρέπει να κοινοποιούνται. Είναι, ε, είναι σημαντικό αυτό και είναι σημαντική η συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και για τις μικρο ε, πιστώσεις. Στη σελίδα 103 αναφέρεται ε, ότι πρέπει να ξεπεράσουμε την αρχή του do no harm, μην κάνουμε βλάβη. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε και με θετικό τρόπο την ε, πολιτική της συνοχής. Νομίζω ότι αυτό εννοείται εδώ. Επίσης ε, θα πρέπει και τα εθνικά κοινοβούλια να κινητοποιηθούν ε, περισσότερο ούτω ώστε να υπάρξει μια επικούρηση και της Κομισιόν. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα εδώ. τέλος, ο ΣΑ έχει καταρτήσει μια διεθνή πλατφόρμα PCD Υπάρχουν προγράμματα της, για να κάνει η Κομισιόν μια παρόμοια πλατφόρμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιες επιτυχίες που να ε, ε, επιδείξουμε ούτως ώστε να δικαιολογηθεί μια τέτοια πλατφόρμα. Ε, σίγουρα χρειάζεται ε, θάρρος, αλλά και από την πλευρά των ε, πολιτικών χρειάζεται όμως να πείσουμε και τους πολίτες για τη ε, χρησιμότητα των προγραμμάτων. Επειδή είναι σύνθετο το θέμα και είναι περιορισμένοι οι πόροι μας, χρειαζόμαστε την πραγματογνωμοσύνη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στην Concord και για το ενδιαφέρον τους. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκέρνς που τον είχε ζητήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή για μια φορά ακόμα να φέρεται σε υπερβολικά πολλά προβλήματα, τα οποία είναι αδύνατο να λύσουμε στο χρόνο που έχουμε. Βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί αναφέρθηκε στο στόχο μας και που υπογράμμισε ποια είναι τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Κοιτάξτε, ως δωρητές πολλές φορές θα πρέπει να κάνουμε ε, μια συνειδητή προσπάθεια να αξιολογήσουμε και τη δική μας δράση. Μήπως δεν λαμβάνουμε υπόψη επαρκώς τις ανάγκες ε, των εταίρων μας, γιατί και αυτό θα ήταν κομμάτι της συνοχής και της συνέπειας. Δεύτερη παρατήρηση. Για την ε, ε, συνέπεια της πολιτικής μας, νομίζω ότι πολλές φορές είμαστε υπερβολικά σεμνοί και κνητρημένοι στην αξιολόγηση που κάνουμε των επιπτώσεων που έχουν οι πολιτικές μας. Θα σας πω πως το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε 10 δις ευρώ ε, στις εξαγωγικές επιστροφές και το 2008 ήταν 300 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είχαμε μια πολύ σημαντική μείωση των εξαγωγικών επιστροφών που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση σήμερα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Και αυτό δεν το τονίζουμε αρκετά. Εντάξει, το 2009 τα πράγματα πήγαν μάλλον άσχημα, προσπαθήσαμε να στηρίξουμε την αγορά γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα όσα έλαβαν χώρα το 2009 έγιναν για να μην πέσουν υπερβολικά οι εξαγωγικές τιμές για το γάλα. Την ώρα που φεύγουμε από την αίθουσα και έρχεται μια άλλη επιτροπή να μας κάνει ερωτήσεις, ε, πάντοτε αισθανόμαστε σαν να είμαστε σε δύσκολη θέση. Στην πραγματικότητα θα, είμαστε, ε, θα έπρεπε να είμαστε πιο πιστικοί για τα όσα κάνουμε και θα ήθελα να ζητήσω από εσάς το εξής. Να δούμε ποια είναι τα ελλείμματα και τα κενά και τα προβλήματα που έχει το σύστημα το δικό μας στην πολιτική ανάπτυξη. Η Γκάνα, για παράδειγμα, για να προστατεύσει την γεωργική της αγορά, η οποία κατέρευε πριν από 10 χρόνια, και αυτό υπό τις επιταγές ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας, να μειώσει, να μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς. Εκεί έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, διαπιστώσαμε πως η Παγκόσμια Τράπεζα έσφαλε. Ενδεχομένως σφάλει και σε αυτή την περίπτωση. Εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής ε, ε, κονδυλίων στην περιοχή αυτή. Και νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το διατυμπανίσουμε και δεν θα πρέπει από σεμνότητα ε, να υποτιμούμε τη δράση μας. Τώρα, για τα εμπορικά θέματα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε μία τεχνική βοήθεια προς όλες τις, αναπτυσσόμενες χώρες για να προετοιμαστούν καλύτερα για το γύρο της Ντόχα. Τελικά με μια εσφαλμένη ε, ανάγνωση της ε, κατάστασης οδήγησε στο να χρειαστεί να υποταχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, στις βουλές κάποιων αναδυόμενων χωρών. Βραζιλία σε παρένθεση χώρες οι οποίες μας επικρίνουν για τη δράση μας. Ενώ αντίθετα πιστεύω ότι χρησιμοποιήθηκαν με πολύ αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τα δικά μας ε, κονδύλια. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε αυτή την αντίφαση. Είμαστε ο μοναδικός δωρητής ο οποίος προσπαθεί πραγματικά να χειραφετήσει τις χώρες εταίρους. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά για το Διεθνές Θεσμικό Σύστημα να σας πω πως η G20 είναι η μεγαλύτερη ασυνέπεια. Εκεί δεν έχουμε εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει μια φοβερή έλλειψη ισορροπίας των απόψεων. Αυτά ήταν τα συμπεράσματά μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, δικές σας προσπάθειες, οι οποίες όπως πάντα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Thank you. Um, I of course agree with lots of the... Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν, να μην τα επαναλάβω. Να ευχαριστήσω και εγώ την Concord για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Οι οι πίνακε είναι πολύ εξυπηρετικοί και μα διευκολύνουν στο σχεδιασμό πολιτική. Όμω, κάποια όρια φαίνεται ότι τα θέτουμε εμεί στον εαυτό μα όταν πρόκειται για την ε, συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Ω Επιτροπή, καλά τα πάμε σε σχέση με άλλε επιτροπέ, αλλά ακόμη και εδώ δεν είμαστε πάντοτε αρκετά συνεπείς. Και να αναφερθώ σε αυτό που μόλις το πρωί συζητήσαμε με τις προφορίες. Κάτι φαίνεται να γίνεται, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο συνεκτικοί. Να λαμβάνουμε υπόψη και το συμφέρον των αναπτυσσόμενων χωρών. Και αυτό να εκφράζεται και στην στάση μας, τη στάση που τηρούμε κατά τις ψηφοφορίες. Πολύ συχνά η Επιτροπή τη Ανάπτυξη ψηφίζει προ μια κατεύθυνση στην Ολομέλεια και όλη η υπόλοιπη Ολομέλεια προ μια διαφορετική. Λόγω χάρη, είχαμε αντιταχθεί στην έκθεση για την ε, συνοχή πολιτικής, ε, της πολιτική πολιτικής την περασμένη φορά. Είχαμε αντιρρήσει σε γεωργικές και αλληλευτικές συμφωνίε. Προσπαθούμε να επηρεάσουμε του συναδέλφου των άλλων επιτροπών, ώστε να συμπαραταχθούν μαζί μα αυτή την, πολιτική, την στάση τη ε, συνοχή. Πάντως νομίζω ότι πολλά μπορούν να βελτιωθούν στις ε, σχέσεις μεταξύ των Επιτροπών και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να δω μια έκθεση για την ε, συνοχή στην αναπτυξική πολιτική. με κάποια συμπεράσματα για τις σχέσεις συνεργασίας που μπορεί να υπάρχουν, για επιτυχή παραδείγματα, για πράγματα που επίσης μπορεί να μην πήγαν καλά ή να μην είναι αρκετά καλά συντονισμένα. Να πούμε δηλαδή ότι αυτή τη μάχη μπορεί να τη χάσαμε. Δεν είμαστε αρκετά συνεκτικοί ακόμα, αλλά το γνωρίζουμε, το συνειδητοποιούμε, ασκούμε κριτική στον εαυτό μα. Γιατί μπορούμε να δούμε λόγω χάρη τα βιοκαύσιμα με μια έκθεση πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εδώ υπήρχε συνεπεί προς προ του στόχου μα για την αναπτυξιακή πολιτική. Επίση, κάτι που θα ήθελα να δω στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη ήταν περισσότερο τεκμηριωμένη με πραγματικά στοιχεία επιχειρηματολογία. Λόγω χάρη ένα πρόσφατο παράδειγμα. Είχαμε την παρουσίαση της μελέτης για τις γενετικούς πόρους και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Και υπόθηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία ότι ε, τα δικαιώματα πολιτική υποκτησίας ε, μειώνουν τη φτώχεια στι αναπτυσσόμενε χώρε. Ενώ βλέπουμε ότι είναι υπέροχα τα δικαιώματα αυτά στην έκθεση τη Επιτροπή για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Κάτι λείπει λοιπόν εδώ. Λείπουν τα αποδεικτικά στοιχεία στον πίνακα. Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και αυτά. Αλλιώ δεν υπάρχει επιχείρημα. Είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι τα πράγματα είναι πολύ όμορφα, όμω ε, κάποιοι μπορούν να τα αμφισβητήσουν. Και εμεί δεν μπορούμε να αντιπαρατάξουμε επιχείρημα. Επιπλέον, για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν αυτό συζητάμε, αλλά αυτό που ήθελα να δω ήταν κάποια αναθεώρηση για το πρόγραμμα εργασίας για την συνοχή. Καλό είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη, αλλά τι απέγινε, ήταν επιτυχές, αποτελεσματικό, τι μαθήματα λύσαμε από την προηγούμενη εφαρμογή του και πώς παρακολουθείτε την ε, εκτέλεση της προηγούμενης έκθεσης ε, για την ε, πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη. Σύντομα θα έχουμε και την επόμενη. Θα έχει το ίδιο περιεχόμενο, γιατί θέλουμε να δούμε τι ήδη έχει υλοποιηθεί, τι πήγε καλά, τι όχι. Λόγω χάρη για τα εστιακά σημεία και τις αντιπροσωπείες, την συνοχή της συνοχής αυτής. Κάποιες χώρες όπως η Πορτογαλία δεν τα έχουν υλοποιήσει ακόμα. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Είναι καλά όλα αυτά για την ε, κατανάλωση τη Επιτροπή και για τις ε, ανάγκες της Επιτροπής, όμως ε, κάπου θέλουμε και εμεί κάποια πράγματα. Έχουμε και εμεί ανάγκε που να ικανοποιηθούμε μια τέτοια έκθεση. Α μην επικαλύπτουμε λοιπόν τι προσπαθίες μα. Νομίζω λοιπόν ότι στην έκθεση τη Επιτροπή μα λείπουν κάποιες κρίσιμες παρατηρήσεις. Στοιχεία που θα μα δείχνουν ξεκάθαρα αν πρόκειται για μια μάχη που μπορεί να χαθεί απλώ. Και καλό είναι να είμαστε ειλικρινεί με του εαυτού μα, γιατί δεν είναι μια απλή διαδικασία η, συνοχή, η πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη. Το γνωρίζουν αυτό οι αρμόδιε υπηρεσίε και το Κοινοβουλίο και τη Επιτροπή. Και κυρίω να βασιζόμαστε σε πραγματικά αποδεκτικά στοιχεία. Είναι σημαντικό αυτό. Η έκθεση τη Concord επίση βοηθά πολύ. Ίσως υπάρχουν κάποιες καλές εδώ ιδέες για τις μελλοντικέ μας δράσεις, αλλά Καλό θα ήταν να μπορούμε να βλέπουμε τι χώρε συνολικά και μία-μία, ώστε να βλέπουμε πώ οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ τι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Γιατί το θέμα είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ λόγου χάρη του γαλακτοκομικού τομέα, που μπορεί να επηρεάζεται από μια συγκεκριμένη πολιτική και να επηρεάζει με τη σειρά του άλλου. Αυτό είναι απλώ μια ιδέα. Επίση, κάτι που θα μα εξυπηρετούσε είναι να δούμε τι επίκειται, όπω ε, η νέα αγροτική πολιτική, η νέα καθεστώτα εμπορικών σχέσεων. Αυτά βεβαίω περιλαμβάνονται και στι μελέτε αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ότι δεν έχει γίνει, καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί. Εάν είναι εφικτό. Θα μα διευκόλυνε. Αυτά. Τώρα. Κυρία Τομπιέσοβα, για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω κάνοντας μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης. Ξέρω πως την έχουμε συζητήσει σε βάθος και γνωρίζουμε το περιεχόμενο, αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια εισαγωγικά. Καταρχήν χαιρετίζω την ανταλλαγή απόψεων και την ευκαιρία να σας κάνω την παρουσίαση που μου δίνετε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση της πολιτικής ε, με συνοχή για την ανάπτυξη και το γεγονό που συζητάτε πτυχέ αυτή τη πολιτική στην Επιτροπή σα μα έχει βοηθήσει πολύ στο παρελθόν και ελπίζουμε πω θα συνεχίσει αυτό και στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση αναμένει με μεγάλη προσδοκία την, ε, με, την ε, γνωμοδότηση ε, του Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα. Το έγγραφο εργασία το οποίο εκδόθηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς, στις 15 Δεκεμβρίου του 2011, είναι η τρίτη έκθεση η σχετική με το θέμα της ε, πόλης οικοχίζων και έχει συνταχθεί με βάση τις δικές σας ε, συνεισφορές αλλά και διάφορες μελέτες. Άρα λοιπόν η έκθεση έχει, ε, βασίζεται, η ποιότητα της εκθέσης βασίζεται και στα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, αλλά και στις συνεισφορές ε, όλων των συντακτών και των άλλων διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε δυστυχώς δεν ε, έχουμε εξετάσει εμείς οι ίδιοι κάθε φορά τις περιπτώσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται καλύπτει τις περιόδους από την προηγούμενη έκθεση του 9 και προσπαθεί να εστιάσει την προσοχή του αναγνώστη σε συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις και στοιχεία. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για μια σφαιρική συνολική έκθεση, αλλά για κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Έχουμε το πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το 2010 και μέχρι το 2013 για το θέμα του PCD και η έκθεση εστιάζεται στα πέντε σημεία κλειδιά που εντοπίστηκαν το 2009 στην έκθεση. Και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε βεβαίως και στο πρόγραμμα εργασία. Έχουμε τα τρία τμήματα της έκθεσης. Το πρώτο είναι τα εγκάρσια θέματα, γενικά εγκάρσια, εφαρμογή των δεσμεύσεων, όπου προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε ποιο αναλαμβάνει ε, τι και ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται. Εκεί επίσης αναφερόμαστε ε, στην τεκμηρίωση ε, του θέματο. και ε, αναφερόμαστε επίσης στα διδάγματα που έχουμε αποκτήσει για τη μεθοδολογία, για τη συλλογή δεδομένων κτλ. Όπως επίσης και να τονίσουμε τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Στο κεφάλαιο αυτό μιλάμε και για την πλατφόρμα για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις και με την ευκαιρία απαντώ και σε μία από τις ερωτήσεις σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στην πλατφόρμα αυτή. Ε, δεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση γιατί παροτρύνουμε τα focal points από τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν και μάλιστα έχει ανοίξει η ε, πλατφόρμα αυτή και για χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη του ΩΣΑ και αυτό μας βοηθάει γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε δύο φορές τις ίδιες συζητήσεις. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν οι εξελίξεις είναι πολύ θετικέ γιατί έγινε μια συνάντηση σε 9 Φεβρουαρίου των Focal Points και Καλέσαμε εκεί και focal points από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο μέλη του ΩΣΑ, που μας επέτρεψε να εξετάσουμε σε βάθος την μεθοδολογία μας. Um, goes also... Στο πρώτο κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, ε, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή την ε, προσέγγιση της, τη μη βλαβερή, το do no harm, γιατί όταν μιλάμε για συνεκτική πολιτική στην ε, ανάπτυξη, ε, συνήθως αναφερόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από τα κακά παραδείγματα. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να αναφερόμαστε και στις συνέργειες ή σε άριστες ε, περιπτώσεις, για να δούμε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει αυτή η πολιτική. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν τις θεωρίες με θετική έκβαση, γιατί η αφήγηση αυτών μπορεί να δημιουργήσει και πολιτική βούληση. Έχουμε τις πέντε ε, ε, περιοχές προτεραιότητας στο επόμενο. Ξέρετε ποιες είναι η ασφάλεια, η μετανάστευση, η εμπορική διάσταση. Δεν θέλω να μπω σε υπερβολικές λεπτομέρειες γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ένα από τα θέματα, για παράδειγμα, και μια από τις επιτυχίες για τις οποίες είμαστε ε, πολύ περήφανοι, είναι η έκθεση αναχώρα, τα προφίλ χωρών. Και η Κονκορδία νομίζω έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Κάποια από αυτά τα οποία δεν παρουσιάζουμε δεν είναι επιτυχίες μεν, αλλά δεν θα τα θεωρούσα και αποτυχίες. Για παράδειγμα, γεωργική πολιτική, αλληλεία. Το γεγονό πω στην προετοιμασία αυτών των πολιτικών θίγονται και κάποιε αναπτυξιακέ διαστάσει ήδη για μα αποτελεί επιτυχία. Δεν θα έπρεπε όμω να βλέπουμε τα πράγματα ασπρόμαυρα, γιατί καμία πολιτική δεν μπορεί να έχει 100% συνέπεια και συνοχή. Άρα λοιπόν ποτέ δεν τελειώνει το έργο μας. Το 3 είναι τα διδάγματα, ο κατάλογος των κρεμωτήτων, τρεχουσών προκλήσεων και προκλήσεων για το μέλλον, συνεισφορά άλλων μερών. Το έγγραφο αυτό δεν παρουσιάζει φιλόδοξες νέες κατευθύνσεις, είναι ένα έγγραφο εργασία της ε, Κομισιόν χωρίς προτάσεις και κατανοώ την απογοήτευσή σα για το ότι δεν έχουμε νέες προτάσεις, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος της συνταξη του κειμένου. Για τη συνέχεια που θα δοθεί, το follow-up, Έχουμε το πρόγραμμα εργασίας που τρέχει μέχρι το 2013. Εκεί έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία πλέον δεν είναι επίκαιρα. Γίνεται μια αξιολόγηση και ετοιμάζουμε και το νέο πρόγραμμα για τη μετά το 13 εποχή. Εκεί είμαστε. Δεν θέλω να σας καθυστερώ. Το έγγραφο είναι προσβάσιμο ελεύθερα στο διαδικτυακό μας τόπο. Θα συζητηθεί στο Συμβούλιο και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι πριν το Φεβρουάριο που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο, συζητιέται ήδη τον Ιανουάριο στο Κοινοβούλιο και αυτό δείχνει πόσο κινητοποιημένοι είστε εσεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. κύριος Γιάγκερσεν. Θα τον παρακαλέσω να είναι σύντομος. Well, thank you. Σας ευχαριστώ. Και εγώ να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Νομίζω είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση για την συνοχή σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχουν ζητήματα συνολικότερα. Μια από τις βασικές μας λοιπόν νέες ιδέες για την συνοχή στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γεωργία να συνεξεταστεί με τι ευρύτερε εμπορικέ σχέσει, εφόσον είμαστε με ένας μεγάλος σε αυτόν τον τομέα. Εδώ η συνοχή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Αλλά η συνοχή ε, είναι κάτι που επιζητούν και οι αναδυόμενες οικονομίε και οι αναπτυσσόμενες χώρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα. Και έχει πολύ αυστηρού νόμου λόγω χάρη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αναπτυξιακή τη πολιτική καθορίζει τις ευρωπαϊκές, εξωτερικές, τις ευρωπαϊκές αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής και δράσης. Αυτές οι πρωτοβουλίες λοιπόν θα πρέπει να είναι και αποτελεσματικέ προκειμένου να προωθήσουμε τις αρχές τις οποίες έχει θεμελιωθεί η Ένωση. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Και κάτι ακόμη. Νομίζω για τα αποδεκτικά στοιχεία που ζητήσατε, η, συνοχή, για την, η πολιτική συνοχή μάλλον για την ανάπτυξη, είναι κάτι που βεβαίω πρέπει να βασίζεται σε αποδεκτικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει κάθε φορά να έχουμε κατά νου ότι είναι και θέμα πολιτική βούληση και προθυμία να υπάρχει πολιτικό διάλογο και να εμπλέκεται και η κοινωνία των πολιτών. Λόγου χάρη, όταν ε, εργαστήκαμε για την κοινή αγροτική πολιτική, συνοργανώσαμε μία συνδιάσκεψη με την ε, ε, με το σύλλογο των Δανών Γεωργών. Ήταν σημαντικό να φουγκραστούμε ότι έχουν να πούν οι Γεωργοί και σε παγκόσμιο επίπεδο και νομίζω ότι αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Γεωργοί. Για μια τέτοια λοιπόν πολιτική κοινή, όπως η κοινή αγροτική πολιτική που έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία 20 χρόνια, είναι σημαντικό να δούμε τι συμβαίνει. Βεβαίω οι επιδράσει δεν είναι οι ίδιε στη Δανία όπω στην ε, Ταϊλάνδη λόγου χάρη, αλλά το θέμα δεν είναι να δούμε μόνο τι γίνεται στι αναπτυσσόμενε χώρε ξεχωριστά και απομονωμένα, αλλά και στην Ευρώπη. Και αυτό πιστεύω ότι και εφικτό είναι και είναι απλό σχετικά, απλώ είναι θέμα πολιτική βούληση και διαλόγου. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Σλίμπερ Γέστραμ για, για το συμπέρασμα. Ευχαριστώ θερμά για όλες ε, τις παρεμβάσεις. Προκύπτει σαφώς ότι σας ενδιαφέρει όλους το θέμα PCD, γιατί είναι σημαντικό δηλαδή το θέμα της βιωσιμότητας των πολιτικών μας. Πολύ δουλειά μας περιμένει. Κύριε Γκέρενς, σίγουρα και έχετε δίκιο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους έγιναν πολλά πράγματα γιατί δεν πρέπει να επικρίνουμε μόνο και να λέμε μόνο τα αρνητικά χωρίς να τονίζουμε και τα θετικά. Αυτό είναι σε βάρος μας. Πιστεύω παρόλα αυτά ότι ο τομέας της συνεργασίας, για παράδειγμα, και με οριακές χώρες αναδυόμενες είναι σημαντικός τομέας. Θα πρέπει να ενταχθούν και εκείνες στις πολιτικές μας. Και πώς θα γίνει αυτό, γιατί δεν έχει νόημα να λειτουργούμε ανταγωνιστικά επί τόπου, ποιος είναι ο καλύτερος δωρητής, ποιος θα κάνει καλύτερα και να επικρίνουμε μόνο τους άλλους, ε, αντί να πούμε ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει ε, ε σύνεση να τα προχωράμε. Μπορούμε να ε, κάνουμε ένα καταμερισμό εργασιών. Πολλή δουλειά λοιπόν έχουμε ακόμη και η Κομισιόν ενδεχομένως κάποια μορφή benchmarking, μια συγκριτική αξιολόγηση θα μπορούσε να δώσει κίνητρα στις διάφορες χώρες, ποιος κάνει τι καλύτερα, ε, ορθές πρακτικές, πώς μπορούμε να τις μιμηθούμε. Σίγουρα υπάρχουν καλά παραδείγματα και νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ε, και θα συμβάλλει και η έκθεση που θα ψηφίσουμε όταν ε, συνεργαστούμε και με τους συναδέλφους από την Γεωργική Επιτροπή και με άλλους ε, για να συνεχιστεί η δραστηριοποίηση στο θέμα αυτό, ε, νομίζω ότι καλό θα είναι. Μπορεί να δουλέψουμε, αλλά δεν βλάπτει. Δίκιο έχετε. Νομίζω σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψε. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Η Συμφωνία της Κοτονόπου, ξέρετε, τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά και το κοινοβούλιο μας ε, καλείται να τοποθετηθεί για αυτήν την Διεθνή Συμφωνία βάσει της σύσταση της ε, δικής μας Επιτροπής. Ο εισηγητή μας είναι ο κ. Κάσμαν, στον οποίο θα δώσω και πάλι το λόγο, για να μας παρουσιάσει εντάχει το όλο θέμα. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο κ. Κάσμαν έχει εξαιρετικού λόγου να θέλει να παρουσιάσει την έκθεσή του αργότερα για λόγους που ακριβώς θα μας εξηγήσει ευθύς αμέσως. Κύριε Κάσμαν, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ευγενικό. Κατά πρώτον, θα πρέπει να παρατηρήσω ευθύ εξ αρχή το κατάφορο λάθο το τίτλο τη έκθεση αυτή στην αγγλική μετάφραση. Διαβάζω second amendment στα αγγλικά, ενώ θα έπρεπε να λέει second revision, δεύτερη αναθεώρηση. Αναθεωρείται η Συμφωνία νου. Βεβαίω, η νομική βάση τη αναθεώρηση είναι το άρθρο 95 τη Συμφωνία και η πρώτη αναθεώρηση ήταν τον Ιούνιο του 2005. Η δεύτερη αναθεώρηση ξεκίνησε το Μάιο του 2009 και οι λόγοι που μα οδήγησαν σε αυτή την απόφαση ήταν πολλοί. Πρώτα απ' όλα, λόγω της πείρας που αποκομίσαμε από την Συμφωνία της Κοτονού και την υλοποίησή της, από την εμπειρία των δράσεων των χωρών και, και του Κοινοβουλίου του ίδιου, ιδίω λόγω τη φύση τη εταιρική σχέση μεταξύ χωρών Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρών ΑΚΕ. Ε, πρέπει να προσαρμοστούμε στι πρόσφατε μείζονε αλλαγέ, στο διεθνέ προσκήνιο και στι σχέσει ε, χωρών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Υπάρχουν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να απτυχθούν προ όφελο των δύο πλευρών, δηλαδή η πολιτική και θεσμική διάσταση, η οικονομική συνεργασία, η περιφερειακή ολοκλήρωση, η ανάπτυξη του εμπορίου, η χρηματοδότηση τη ε, συνεργασία, το προγραμματισμό, η δημόσια διαχείριση και τα σημαντικά ζητήματα των, σχέσεων, συμφωνιών εταιρική σχέσης και οι συνέπειέ τους. Οι Όπως θυμούνται τα μέλη της Επιτροπής, επαναδιαπραγματευτήκαμε σε αυτούς τους όρους την συμφωνία της Κοτονού, το, την επέγραψε στο Συμβούλιο, την κύρωσαν τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του και το Κοινοβούλιο. Έχω παρακολουθήσει στενά το θέμα και κατά καιρού αισθάνθηκα και ανυπομονησία προ τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων. Αλλά υπό την Ισπανική Προεδρία στο Συμβούλιο αποφασίστηκε τελικά να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση και από την πλευρά του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ε, επικρίνω τον Επίτροπο. Όμω για κάποια ζητήματα που δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση, όπω τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη διακριτική μεταχείριση βάσει των διαφορών, εκεί υπήρξαν ε, υπαναχωρήσει. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι όπου η χώρα ΣΑΚΕ αντιστάθηκαν στη στάση που τηρήσε ο Επιτροπό μα και η διαπραγματευτική μα ομάδα. Βεβαίω, εάν υπαναχωρήσουμε μπροστά στην τεράστια σημασία της, ε, του μη διαπραγματεύσιμου, της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ουσιαστικά ε, είναι σαν να λέμε ότι τα πράγματα αυτά είναι διαπραγματεύσιμα τα δικαιώματα αυτά και να τα διαπραγματευόμαστε μπορούμε και να τα αγνοούμε ενδεχομένω. Δηλαδή να τα αποκλείουμε και από διεθνεί συμφωνίε. Αυτό νομίζω και εγώ προσωπικώ και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Δεν μπορούμε να συγκατανε... συγκατατεθούμε. Άλλωστε και στην έκθεση της κυρίας Ζολή από τον Δεκέμβριο του 2009 εντοπίζεται το στοιχείο αυτό. Τα περισσότερα λοιπόν από τα σημεία που εντοπίζει η κυρία Ζολή δεν καλύπτονται από το τελικό κείμενο. Νομίζω λοιπόν, όπως έχει ήδη εκφράσει με ψηφίσματά της η Επιτροπή μας και ως προς τις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο άρθρο 8.4. Μη διακριτική μεταχείριση και η κάλυψή τη, η προστασία δηλαδή, η αποφυγή τη να συμπεριλαμβάνονται στο πολιτικό διάλογο. Όπως ορίζει και η διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την πλευρά των χωρών ΑΚΕ, άλλωστε, υπήρξαν και αντιστάσει ω προ τη συμπερίληψη τη ε, της μεταχείριση μεταχείρισης βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού. Εάν υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τη συζήτηση των θεμάτων αυτών, δεν θα ήταν μείζονο σημασία το θέμα, εάν η ομοφιλοφιλία δεν ε, ήταν ένα σοβαρό έγκλημα που πολλές φορές τιμωρείται αυστηρά σε πολλές από τις χώρες, τις, ε, τις χώρες ΑΚΕ. Δεν μπορούν λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστέλουν το μήνυμα ότι δεν διατηρούν στεναρές ε, στεναρές τάσεις στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη μη διακριτική μεταχείριση και κυρίω στο ζήτημα αυτό που δεν ήθελαν καθόλου να διαπραγματευτούν οι χώρε ΑΚΕ για το σεξουαλικό προσανατολισμό. Το να τηρήσουμε τη σιωπή ουσιαστικά είναι σαν να αφήνουμε στη μέση τον κάτι που έγινε στη δεκαετία του 80 με τον πόλεμο κατά του AIDS από τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μας οδηγήσει σε θάνατο. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Δεν θέλω λοιπόν εγώ να έχω ε, συγκατατεθεί σε μια τέτοιου είδους πολιτική απόφαση. Ιδάλλως ε, αντιφάσκουμε με όσα έχουμε υποστηρίξει από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Επίσης αναφέρθηκαν και άλλες ανησυχίες για να μεταπεράσω λίγο από το θέμα που ίσως αναφέρω πολύ συχνά για την ε, καλή διάθεση κάποιων μελών της Επιτροπής. Θέματα που αφορούν την ε, απουσία αναφοράς στο ισότιμο εμπόριο, το δίκαιο εμπόριο, την πρόθεση των μικροπιστώσεων για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Επίσης, διερωτήθηκα και δεδομένη της παρουσίας της Επιτροπής, εάν μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί η λισαβονοποίηση της συμφωνίας όπω είχε αναγγείλει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τελικά δεν περιλαμβάνεται στην τελική εκδοχή του κειμένου αυτή που έχουμε μπροστά μα. Πώ θα προχωρήσουμε λοιπόν. Όπω είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τι δικέ μα ανησυχίε και κανονικά είναι πρόθυμη να τη συζητήσει μαζί μα. Ο Επίτροπο Πίμπαλξ έχει επικοινωνήσει μαζί μου υπό την ιδιότητά μου ω εισηγητού και συμφωνήσαμε να οργανώσουμε μια εκδήλωση για το θέμα τη μη διακριτική συμπεριφορά εντό τη συμφωνία αυτό είναι μια εξαιρετική ευκαιρία κατά την άποψή μου να συζητήσουμε πράγματα που κάποιοι θα ήθελαν να τα αποσκοπήσουν και ενδεχομένω να καταλήξουμε σε κοινή συνεννόηση ή κοινού στόχου. Θα οργανωθεί του ερχόμενου μήνε η εκδήλωση αυτή και αυτό είναι ένα βήμα μια κοινή καλή θέληση από την πλευρά τη Επιτροπή και του ίδιου του Επιτρόπου. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να περιμένουμε τι συζητήσει που θα γίνουν ε, εντό Επιτροπή ε, σε συνεργασία με τους πρέσβεις των χωρών και τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη του Συμβουλίου που θα προσκληθούν στην εκδήλωση αυτή. Οπότε θα ήθελα να περιμένουμε και την ε, διεξαγωγή της εκδήλωσης αυτής πριν ε, δώσω την τελική μορφή στην έκθεσή μου. Θα ήθελα επίσης να τονίσω, εφόσον έχω και τη συμφωνία των συναδέλφων, ε, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είμαστε, και το τονίζω αυτό, δεν είμαστε διατεθειμένοι να προκαλέσουμε την ομοιρία του ή ουδήποτε εφόσον δεν επηρεάζονται οι οικονομικέ ρήτρε τη Συμφωνία Κοτονού. Υπάρχει και δυνατότητα τρίτη αναθεώρηση το 2015, εφόσον χρειαστεί, πριν εκπνεύσει η Συμφωνία το 2020. Το Κοινοβούλιο, όπω έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, και όπω είπα και εκ μέρου του κ. Μπέρμαν σήμερα το πρωί, λαμβάνει πολύ σοβαρά τον ρόλο που του έχει ανατεθεί. Ιδίω ω προ τη διαδικασία τη συνένεση. Για το σκοπό αυτό, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε τι συζητήσει που θα προκύψουν και θα προκαλέσει αυτή η εκδήλωση και με τον δέοντα σεβασμό και την δέουσα προσοχή να προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρος, να δώσουμε το λόγο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Γκέρενς που έχει μια ερώτηση. Οπότε κατάλαβα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κάσμαν για τη συνοπτική εικόνα που μας παρουσίασε για τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού. Όντως, γνωρίζει το θέμα πολύ καλά Απλώς στα σημεία που εντόπισε και ο Μάικλ για το θέμα της μη διακριτικής συμπεριφοράς. Είχα ένα μακροσκελή συζήτηση με τον Επιτροπό Πίμπαλξ και όντω έχει ακουστεί η ιδέα να διοργανωθεί μια ημερίδα, μια πρωτοβουλία για να το συζητήσουμε αυτό περαιτέρω. Επίση, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αντίσταση από την πλευρά των χρόνων και τα θέματα αυτά να συζητηθούν λεπτομερέστερα. Το είδατε και στη μεικτή, την, ισοβαρή, ισομερή μάλλον ε, διάσκεψη. Το είδατε και τις, τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις της διάσκεψης αυτής. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι όντω αλήθεια ότι σε κάποιες χώρες ο σεξουαλικό προσανατολισμό, ιδίω η ομοφιλοφιλία, είναι ποινικά κολάσιμο συμπεριφορά. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να τηρήσουμε μια στάση αμετακίνητη. Τέτοιου είδους νομοθετικά μέτρα έχει ζητηθεί να ανακληθούν όπως στη Ρουάντα, στο Μπουρούντι, στο Μαλάουι Αυτή τη στιγμή νομίζω να προβλήματα υπάρχουν στον Ήρα. Παλιότερα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προσώπων μα και τη ύπαρξη εκπροσώπου ε, εντόπισαν τα θέματα αυτά στι ε, ενδιαφερόμενε χώρε και του είπαν ότι το να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να μην καταστούν ε, και νέες στι τις πολιτικές που διοργανώνουμε από κοινό με τι χώρε εκεί. δεν είπαμε να περάσουμε και σε πλήρη απαρίθμηση των περιπτώσεων μη διακριτική μεταχείριση όπω γίνεται και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Για τι υπόλοιπε πτυχέ, για την απουσία τη λισαβονοποίηση. Τη στιγμή που υπογράφει η συμφωνία στο Ουάγκα του Γκου, η, συμφωνία, η συνθήκη της Λισαβόνας δεν είχε τεθεί ακόμη σε ισχύ. Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοινοποιούσε στις χώρες ΑΚΕ τις αλλαγές που θα προκαλούσε η θέση σε ισχύ της συνθήκης τη Λισαβόνα. Δηλαδή, η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο, στο Κοινό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Μεικτό Συμβούλιο των Πρέσβων για την ώρα έχει αποστείλει επιστολή η Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτει το σχέδιο συμφωνίας που έχετε μπροστά σας και το οποίο πρόκειται να εγκριθεί. Επιστολή η οποία τελικά ανακλήθηκε από το Συμβούλιο. Θεωρήθηκε ότι υπήρχαν ζητήματα εκκρεμή ακόμη ω προς την εκπροσώπηση την εξωτερική εκπροσώπηση τη Ένωση. Ξέρετε ότι η Λισαβόνα τελικά δεν απλούστευσε τα πράγματα από αυτή τη σκοπιά. Εδώ λοιπόν Απομένουν στοιχεία τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν. Πάντω, μεταξύ των προθέσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να υποβάλει στην κρίση σα σύντομα αυτή την επιστολή, ώστε να διευθετηθούν τα θεσμικά ζητήματα που, προκαλεί προκύπτουν από τη Συμφωνία Κοτονού και σύμφωνα με τι διατάξει τη Συνθήκης τη Λισαβόνα. Επειδή πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, θα σταματήσω νομίζω εδώ. Και σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να συζητήσει τα υπόλοιπα σημεία που ενδιαφέρουν τον εισηγητή. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία να οργανωθεί κοινό διάλογο με τον Επιτροπό Πίμπαλξ θα μπορούσε να μα οδηγήσει σε συμπεράσματα θετικά και επικοδομητικά για την ετοιμασία τη τελική έκθεση από την Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Πρόεδρο, κύριε Γκέρεν, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι στο πλαίσιο της συζήτηση αυτής δεν μπορούμε να αποφύγουμε μια αλήθεια η οποία υποκρύπτεται καθ' τη διάρκεια της συζήτησής μας. Η Κοτονού απειλείται με διάλυση, είτε το θέλουμε είτε όχι, με τις διμερείς περιφερειακές συμφωνίες. Η συνοχή μπορεί τελικά να πληγεί στην ίδια την καρδιά της, την καρδιά του θέματος. Και ως προς το σχόλιο του Μάικλ, θέλουμε να ακουστούν οι διεκδικήσει του Μάικλ. Θα πρέπει να τον στηρίξουμε σε αυτόν τον δρόμο. Και πρέπει το πλαίσιο αυτό, το ενιαίο πλαίσιο να παραμείνει. Ο χώρος, ο ενιαίος χώρος αξιών να παραμείνει αδιάρρητος. Νομίζω, το συζητήσαμε το θέμα αυτό με κάποιον που γνώριζε πολύ καλά του σχετικού προβληματισμού. Χωρί τη σφαιρική προσέγγιση με όλε τι χώρε ΑΚΕ, δεν θα καταφέρναμε ποτέ να έχουμε αυτή τη συμφωνία. Εάν είχαμε αρχίσει να. Αν δεν είχαμε ξεκινήσει από τα διαφορετικά στοιχεία που μα διακρίνουν, δεν θα είχαμε καταφέρει ποτέ να συνθέσουμε αυτό το τελικό δημιούργημα που θυμίζει μοσαϊκό. Εάν λοιπόν δεν έχουμε την Κοτονού, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά το 2020 στην πραγματικότητα. Στην ε, Κοτονού ελήφθησαν σοβαρέ αποφάσεις που πάνε και μακριά. Τι γίνεται με τη γενιά των νέων ε, συμφωνιών. Νομίζω ότι ο ιδιωτικό τομέα δεν τα πολύ καταφέρνει. Μετά το Βερολίνο δεν προχωρήσαμε και πάρα πολύ. Και επίσης κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Η εκόλευση τη κοινωνία των πολιτών δεν είναι κάτι που μα έχει ικανοποιήσει ω τώρα. Ίσως την δημοσιονομική μας στήριξη θα πρέπει να πετήσουμε ισχυρότερε πολιτικέ ω προ την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να στηρίξουμε τι κοινωνίε των πολιτών στι χώρε αυτέ. Διότι θα πρέπει οι πολίτε να αναλάβουν και νέε ευθύνε. Πολλαπλασιάζονται οι ευθύνε του, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητέ του, αυτέ που προκύπτουν από την οργάνωση του κράτου. Άρα, δεν θα θέλαμε να θυσιαστεί η Συμφωνία ο Κοτονού στο βωμό τη Αφρικανική Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε την ε, κατάλληλη ισορροπία ώστε να ε, συνδυάσουμε τα καλύτερα στοιχεία και των δύο. Και να βελτιώσουμε τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Διότι μετά στην Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Τελικά δεν έχουμε καταλάβει ποιο κάνει τι. Εάν δει κανεί τα ανακοινοθέντα όσων συμμετείχαν, μπορεί να εντοπίσει κάποια στοιχεία, αλλά οι περισσότεροι συσσωρεύουν απορίε, στι οποίε δύσκολα βρίσκουν απαντήσει. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον Τζάρλς για τα σχόλια που έκανε γιατί όπως πάντα ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα και έθιξαν και τον πυρήνα των όσων μας αφορούν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχω συστήσει ένα ίδρυμα για την κοινωνική δικαιοσύνη ε, για τους ομοφιλόφιλους και τις ομοφιλόφιλες και καταφέραμε να, νι... καταφέραμε να αλλάξουμε την προσέγγιση ε, που ακολουθούσε η κυβέρνηση με τη βοήθεια του ιδιωτικού ε, κλάδου. Ε, γιατί ε, μπορούμε να διδαχτούμε από τι άριστε πρακτικές και νομίζω ότι θα πρέπει ε, αυτό το δίδαγμα ε, να το χωνέψουμε. Χρησιμοποιώ το Google σε διεθνέ επίπεδο και έχουν μία μονάδα για τη διαφορετικότητα και εκεί που βρίσκονται, στις χώρες που βρίσκονται, εξασφαλίζουν να μην γίνονται διακρίσεις και η διαφορετικότητα να προωθείται από την ίδια την εταιρεία σε χώρες όπω οι χώρε ΑΚΕ. Άρα λοιπόν ο ιδιωτικός κλάδος είναι ένας εξαιρετικός μηχανισμός και συμφωνώ με τα όσα είπες Ντομινίκ και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη αρμοστία η οποία ε, έχει λάβει μια πολύ στεναρή στάση ε, εναντίον οποιασδήποτε διάκρισης ε, είτε είναι φιλετική, είτε σεξουαλική, είτε κάποια άλλη. Θα ήθελα αν μου κάνετε τη χάρη για ένα λεπτό να μιλήσω για τα τελικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεών μας. Ε, ανάμεσα σε άλλο, ο διάλογος θα εστιαστεί σε θέματα που μας ανησυχούν όλους και οι χώρες ΑΚΕ μπορούν να μας πούν εντάξει δεν είναι θέμα αμοιβές ανησυχίες, με το συζητήσουμε. Αλλά είναι θέματα που βοηθούν στη γενικότερη επιτυχία της συμφωνίας. Για παράδειγμα, ε, υπερβολικές δαπάνες στρατιωτικές, ε, παιδική δουλεία, ε, διακρίσεις για οποιοδήποτε ε, λόγο, ε, λατρεμπόριο όπλων, όλα αυτά. Και όταν μιλάμε για διακρίσεις, μιλάμε για τον περιφρονητικό όρο άλλης ταυτότητας, άλλης κατάστασης, το other status που λέμε στα αγγλικά. Εάν λοιπόν δεν αναγνωρίζεται η κατάσταση κάποιου από, την, από κάποια χώρα και τότε δεν μπορούμε να συζητήσουμε καν τα θέματα μη διάκρισης, εκτός βεβαίως ε, εάν έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Ντομινίκ, Ευχαριστώ που αναφέρθηκες στην Ρουάντα. Στην Ουγκάντα είδαμε πως έγινε μια προσπάθεια να εξαχθεί αυτό, αυτή η νομοθετική πράξη ε, μίσους κατά των ομοφιλοφίλων. Η Ρουάντα το πέρασε από το κοινοβούλιο και κατέληξε στο εξή συμπέρασμα πως η ιδιωτική ζωή των πολιτών ενδιαφέρουν μόνο τους πολίτες. Και η Ρουάντα θα ακολουθήσει την αρχή της μη διάκρισης και δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους νομοθετήματα. Ρουάντα. Ένα φάρος ελπίδας και νομίζω πια και η Τζαμάικα. Έχουν εκλέξει ένα νέο πρωθυπουργό, ο οποίος είπε πως θα καταργήσει την απαγόρευση για τις λεσβίες ε, και τους ομοφιλόφιλους ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η νέα Πρωθυπουργό ε, θα καταργήσει αυτή τη διάκριση για το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά θα κάνει και δημοψήφισμα για να καταργήσει αυτά τα φρικτά απομεινάρια του ε, απεικιοκρατικού βρετανικού ε, δικαίου που κάνουν διακρίσει κατά των ομοφιλοφίλων. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν, κάνουμε, όταν σημειώνουμε πρόοδο, σημειώνουμε πρόοδο γιατί κάποιοι έδρασαν με θάρρο και δεν εκρύφθηκαν πίσω από το δάχτυλό του όπω κάνουν κάποιοι που με διάφορε προφάσει προσπαθούν να του αποτρέψουν από το να κάνουν το καθήκον του. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο το συμπέρασμα. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο 17 η Επιτροπή μας έστειλε μία αντιπροσωπεία στη συνάντηση που έγινε στο Μπουσάν από 29 Νοεμβρίου μέχρι 1 Δεκεμβρίου, όπου πάνω από 3.000 σύνεδροι εξέτασαν την πρόοδο στην εφαρμογή των αρχών της δήλωσης του Παρισιού και για να συζητήσουν πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την αποδοτικότητα της ε, ε, ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακής βοήθειας ε, στα πλαίσια μιας ανάπτυξης που βρίσκεται σε συνεχή μεταλλαγή. Η υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης στο Μπουσάν μεταξύ των Υπουργών των αναδυόμενων των Αναπτυσσόμενων και των Αναπτυγμένων χωρών μιλάμε για ε, μια τριγωνική σχέση με την κοινωνία των πολιτών και με την συνεργασία ε, νότου-νότου ε, μας οδήγησαν στο να συζητήσουμε σήμερα τα αποτελέσματα που ακολούθησαν από τις διαπραγματεύσεις την ομάδα των ΣΕΡΠΑ που είχαμε τον κύριο Γουστάβο Μάρτιν Πράντα που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω πρώτα απ' όλα βέβαια στην επικεφαλής της αντιπροσωπής αυτής την κυρία Κέλλερ το λόγο για να μας εξηγήσει

Πάνω από 3.000 σύνεδροι ήταν, ήταν μια, τεράστια εκδήλωση, ε, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, υπουργοί κλπ. Πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών παρευρέθησαν μεταξύ άλλων. Για πρώτη φορά ήταν επίσημη αυτή η ε, εκδήλωση των εμπλεκομένων και συμμετείχαμε στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ στις 29 Νοεμβρίου το Κοινοβουλευτικό Φόρουμ προφανώς, ε, με συμμετοχή από βουλευτές ε, από όλο τον κόσμο. Είχαμε ε, πάει επίσης και στο προηγούμενο που ήταν για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, ενδιαφέρουσα εμπειρία και έγιναν και διμερείς συναντήσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα, με την Concord, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Είχαμε και διμερείς με τον Επίτροπο Πίμπαλξ. Χαιρόμαστε για την πρόοδο σχετικά με την ατζέντα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και υπήρξε μεγαλύτερη δέσμευση για τη δημοκρατική διοκτησία και τη βοήθεια ε, και είναι σημαντικό και η Κίνα και άλλοι που ήταν το θέμα αν θα έμπαιναν ή όχι τελικά προσχώρησαν μετά από πολύ ε, διπλωματία και ε, διάφορες κινήσεις και λίγμους. Ήρθαν λοιπόν στο τέλος. Έχουμε λοιπόν τώρα ε, ενισχυμένη ε, δέσμευση για μεγαλύτερη διοκτησία σε σχέση με την βοήθεια, συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τον επιμερισμό της βοήθειας και την εκτίμηση του αντίκτυπου που θα έχει Επίσης ε, έχουμε την αυξημένη χρήση συστημάτων ε, αναχώρα, και όχι ε, συνολικά και ε, καλύτερη διαδικασία εξασφάλισης αποτελεσματικότητας. Και ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών με εκπροσώπους συμμετείχαν ε, για να υπάρχει σωστή εστίαση. Επίσης ένα σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε εκεί είναι ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είπαν ότι θα ε, προσχωρήσουν στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια και αυτό ήταν πολύ θετικό. Ήταν κάτι που αναδείχθηκε, ελήψη άλλων ίσως θα έλεγε κανείς. Τώρα κάτι αρνητικό Είχαμε την τελική διακήρυξη όλων, ένα κάπως κείμενο αφηγηματικό, χωρίς πολλές δεσμεύσεις ή δείκτες που θα λένε ότι αυτός είναι ο στόχος μας και αν συμβούν αυτά και εκείνα θα θεωρήσουμε ότι επετεύχθη. Την τελευταία στιγμή υπήρξαν κάποια καυτά θέματα που ε, συμπεριελήφθησαν. Τελευταία στιγμή η προσέγγιση βάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτέλεσε ένα επίμαχο θέμα και τέλος αυτή η συνολική εταιρική σχέση για τη συνεργασία για την ανάπτυξη που είναι μια παγκόσμια δράση αν θέλετε που θα αντικαταστήσει και του ΩΣΑ την αντίστοιχη ε, πολιτική. Βέβαια δεν ξέρουμε απόλυτα τι θα είναι αυτό το καινούριο εις ό,τι αφορά τη δομή του γιατί υπήρχαν ε, πολλοί που ήταν κατά των νέων δομών, τι θα κάνει, τι αρμοδιότητες θα έχει και ποιος θα είναι μέλος, αν μπορεί κάποιος να προσχωρήσει ως μέλος. Όλα αυτά τα θέματα δεν, ήταν, δεν έχουν αποσαφινιστεί ακόμα. Επίσης ε, ακούσαμε από τον Επίτροπο Πίμπαλς ότι δεν θεωρεί ότι αυτό είναι ε, κύριο για την απτυξιακή ατζέντα. Ε, έχουμε τις ε, δεσμεύσεις ε, των Παρισίων και της Άκρα που υπάρχουν, αλλά όταν έρχονται και σε μια συνεδρίαση 3.000 άνθρωποι μπορεί να θέλει κανείς να δουλέψει περισσότερο πάνω στους στόχους και να επιφέρει και κάποιες τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προηγούμενα τέτοια φόρουμ ψηλού επίπεδου ήταν, είχαν, είχε πρωτοπόρο ρόλο. Ε, αυτό διαφοροποιήθηκε λίγο. Οι άλλες αναδυόμενες χώρες ήταν επίσης μεγάλοι παίκτες, ε, παράγοντες και δεν ήταν ο ηγετικό ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δηλαδή τα κράτη-μέλη ήταν στο προσκήνιο, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κρίμα όμως. Θα έπρεπε όλοι να είναι ενωμένοι σε, αυτό το, σε αυτά τα θέματα. Επίσης η αντιπροσωπεία δεν προσεκλήθη στη συναντήσει συντονισμού, αν και ζητήσαμε, είχαμε ζητήσει από πριν να προσκληθούμε. Δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο. Και δεν ήταν και πολύ ευγενικό το μήνυμα που δεχτήκαμε. Θα δούμε την επόμενη φορά τι θα γίνει στην επόμενη προεδρία. Μπορεί όμως και να μην γίνει άλλο. Ε, μπορεί να μην υπάρξουν ε, τέτοιες ε, υψηλού επίπεδου διασκέψεις για την αποτελεσματικότητα τη βοήθεια. Επίσης, μέσα αυτή τη χρονιά ε, θα υπάρξουν πιο συγκεκριμένοι δείκτες σαν ορόσημα, αν θέλετε, για τη μέτρηση των επιτυχιών μας. Και η διαμόρφωση αυτών των δικτών και των οροσίμων θα είναι πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί θα μπορούμε να τους παρακολουθούμε και να τους επηρεάζουμε. Αφού διαμορφωθούν, μετά θα πρέπει να τηρούνται και να παρακολουθούνται. Ευχαριστώ. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να συμφωνήσει και η κυρία Θεοχάρου με αυτά που είπα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κέλλερ. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η έκθεση. Νομίζω θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαρτίν Πράδα πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα. Νομίζω ότι πολύ σωστά εξήγησε η κυρία Κέλλερ αυτό το φόρουμ στην Μπούσαν υψηλού επίπεδου. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Ήταν μια εκδήλωση η οποία σίγουρα θα επηρεάσει το πρόγραμμα ε, σε θέματα αποδοτικότητας αντεξιακής βοήθειας για πολλά χρόνια. Ήμουν ο Σέρπα, ο οδηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ιχνηλάτης, ε, στην ε, Νότιο Κορέα και θα ήθελα να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις, κυρίως για τα αποτελέσματα του φόρου, μια και πιστεύουμε πως ε, πρόκειται για μια ξεκάθαρη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν να υπογραμμίσω τον εξαιρετικό συντονισμό που είχαμε μέχρι τον Μπούσαν και, στο ίδιο, και στην ίδια την πόλη αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Στις ε, συναντήσεις των ΣΕΡΠΑ είχαμε τρία κράτη-μέλη, ε, που εκπροσωπήθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε και νομίζω πως τα πήγαμε θαυμάσια και στο συντονισμό και στην παρουσίαση της θέσης Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όπου ομόφωνα στήριξαμε τις ίδιες θέσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο και από τα αποτελέσματα, γιατί φαίνεται ότι πολλά από τα θέματα τα οποία υπέβαλε πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά το Συμβούλιο, μια και στους στόχους του Συμβουλίου είχαμε ε, τα αποτελέσματα ε, της ε, πόλης Μπούσαν, ε, νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε ικανοποιημένοι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά παράλληλα να σα πω πως είχαμε και μεγαλύτερη εμπλοκή στο φόρουμ αυτό από πλευρά τη κοινωνία των πολιτών και στην ίδια την ομάδα των ΣΕΡΠΑ αλλά όπως επίσης και του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο και σίγουρα βελτίωσε ε, την ε, σφαιρικότητα των αποτελεσμάτων. Έχουμε πολύ ξεκάθαρους στόχους σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επί της ουσίας και επί των διαδικασιών. Θεωρούμε λοιπόν πως τα έγγραφα τα οποία προέκυψαν ε, αντανακλούν με ιδιαίτερη επιτυχία τα στοιχεία αυτά. Σε κάποιους χώρους που ήθελε να χρησιμοποιήσει το φόρουμ της Μπουσάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τονίσει τη σημαντική προόδο που κάνουμε στο να είμαστε αποδοτικοί, Πρέπει να σας πω πως πρώτα στον κοινό προγραμματισμό που ήταν το βασικό θέμα και το δεύτερο βασικό που ήταν η διαφάνεια, ε, τονίστηκαν ικανοποιητικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης ε, και στο κύριο τμήμα και στις συνοδευτικές εκδηλώσεις αλλά και στα ε, έγγραφα συμπερασμάτων. Συμφωνούμε απόλυτα με την κυρία Κέλλερ. Ένα από του βασικού στόχου τη πόλη αυτή, τη Μπουσάν, δεν ήταν μόνο να επιβεβαιώσει και να την ε, δέσμευση που έχουμε αναλάβει και στο Παρίσι και στην Άκρα, αλλά όχι μόνο να εξασφαλίσει πως οι δεσμεύσεις αυτές θα ολοκληρωθούν και θα ε, εκπληρωθούν με μεγαλύτερη πληρότητα στο μέλλον, αλλά πως και προοδευτικά θα αναλυφθούν και από την πλευρά των αναδυόμενων δωρητών. Τμήμα των συζητήσεων στην Πουσάν και μέχρι την Πουσάν ήταν το πώς χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία μπορούν να μας συνοδέψουν στις προσπάθειές μας, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και θα είμαι ειλικρινής. Το αποτέλεσμα εκεί πολύ απέχει από το να δεχτούν οι χώρες αυτές τις αρχές και τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλάβαμε στο Παρίσι και την Άκρα partnership uh, τους ζητήσαμε να συμμετέχουν σε αυτήν την εταιρική σχέση και όσο μπορούν να εγκρίνουν και να υιοθετούν τις αρχές αυτές τις δικές τους προσπάθειες συνεργασίας και ε, βοήθειας. Βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της διαδρομής, δύσκολα το δέχτηκαν και είναι σαφέστατο πως μόνο μέσω μιας αποδοτικής και νέας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να λάβουμε απτά αποτελέσματα. Τώρα, πώς θα είναι αυτή η εταιρική σχέση. Το λέει και το έγγραφο που προέκυψε. Ξεκινά αυτή τη στιγμή να τρέχει μια εξάμεινη διαδικασία συζητήσεων σε μια ομάδα η οποία θα είναι παρόμοια, αλλά μάλλον διευρυμένη σε σχέση με την ομάδα των Σέρπα που προετοίμασαν ε, την Μπουσάν και εκεί θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες αποκρίσεις στην ερώτηση το ποιος θα συμμετέχει στην παγκόσμια εταιρική σχέση, ποιοι είναι οι δείκτες που θα πρέπει να εκπονηθούν και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε ε, την εκπλήρωση των ε, δεσμεύσεων, ε, των προηγούμενων και των μελλοντικών δεσμεύσεων και προφανώς το ποια θα είναι η διαδραστική σχέση μεταξύ των πιο τεχνικών συζητήσεων και του υπουργικού επίπεδου, όπως είχαμε στην Πούσαν. Όντως, συνήθως ο ήταν ε, ο οικοδεσπότης αυτών των εργαστηρίων για την αποδοτικότητα και ε, έχει δημιουργηθεί μια σειρά επικουρικών ε, δομών, κατά τη γνώμη ορισμένων, ένας, μια υπερβολική πληθώρα δομών, οργανισμών και σωμάτων. Εκεί χρειάζεται να εξορθολογήσουμε και να μεταφερθούμε από το παγκόσμιο επίπεδο το οποίο οδηγείται από το όσα συμβαίνουν στο Παρίσι σε ένα ε, επίπεδο εθνικό ε, και νομίζω ότι για ε, την παγκόσμια εταιρική σχέση αυτή θα υποκαταστήσει τις προηγούμενες δομές και την ομάδα εργασίας και επαναλαμβάνω θα είναι πιο ανοιχτή με μεγαλύτερη συμμετοχή Κίνα, Βραζιλία κλπ. Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα και πάλι ε, βρισκόμαστε στην ε, αφετηρία μιας διαδικασίας για να ε, καταφέρουμε να συνταχθούν μαζί μας οι αναδυόμενοι δωρητές. Τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στηριχθούν, όπως επίσης και τα συμφέροντα των χωρών εταίρων μας, γιατί όλοι συμφωνούμε στις αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας η μόνη μου αντίρρηση στα όσα είπε η κυρία Κέλλερ ήταν η, κατά πόσο ήταν ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πουσάν. Κατά τη γνώμη μου έγινε εξαιρετικό συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και αυτό άλλωστε απηχείται στις δύο παρεμβάσεις που έγιναν σε υπουργικό, επίπεδο, σε υπουργικό επίπεδο στην Πούσαν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, καταληκτική συνάντηση αλλά και στο γεύμα του Υπουργικό, όπου ο Επίτροπος Πίβαλ πήρε το λόγο εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιο από τα κράτη-μέλη. Μίλησε επίση. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Θεοχάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με την κυρία Κέλλερ. Θα συμφωνήσω επίσης ότι σίγουρα τον Μπουζάν θα επηρεάσει στο μέλλον τις εξελίξεις, αλλά δεν ξέρω αν θα το επηρεάσει αποτελεσματικά, πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η επιρροή που θα έχει στην παραπέρα βοήθεια. Δεν έχει ξεκαθαρίσει επίσης ακόμη αν ήμασταν εκεί ως παρατηρητές, δηλαδή το στάτους των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπαν ότι ήμασταν ως παρατηρητές, εγώ δεν αντελήφθηκα ότι ούτε καν αυτό είχε διασφαλιστεί. Η απουσία των εκπροσώπων των κρατών μελών ήταν επίσης ένα αρνητικό στοιχείο. Βεβαίω η Επιτροπή είχε εξαιρετική παρουσία, δεν μπορούμε να είμαστε επικριτικοί σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τις συζητήσεις αυτές καθεαυτές, αναλύθηκαν όλοι οι φαύλοι κύκλοι της αναποτελεσματικότητας της βοήθειας. Βρέθηκαν όλα τα σημεία στα οποία δεν, είναι, δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, όλα τα αρνητικά, συζητήσαμε με την κοινωνία των πολιτών, αλλά δυστυχώ αυτό που αντελήφθηκα ήταν αυτοί που ήθελαν, η, κοινωνία των πολιτών βασικά εκπροσωπείται από αυτού που ήθελαν να διαχειριστούν τη βοήθεια και όχι τόσο πολύ από αυτού που θα μπορούσαν να δεχτούν την ε, βοήθεια, αλλά δεν ετέθηκε εκείνη η γραμμή που θα βοηθήσει δραματικά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας. Δηλαδή όλα παραπέμπονται σε κάποιες δορυφόρες συνελεύσεις, σε κάποιες δορυφόρες, δορυφόρα σεμινάρια και συγκεντρώσεις και συμφωνίες που πραγματικά αν μείνουμε σε αυτό το μοντέλο που υπήρχε μέχρι τώρα χωρίς να βελτιωθεί, όπως είπε η κυρία Κέλλερ, και το ζήτημα της δημοκρατίας, σίγουρα θα παραμείνουμε στα ίδια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Γκέρεντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία πράγματα έχω να πω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την κυρία Κέλλερ που έκανε πολύ, έτοιμασε μια πολύ καλή έκθεση για τη συμμετοχή της ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου και εκπρόσωπος στο Ουζάν. Έπειτα, νομίζω πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για το γεγονό ότι οι αναδυόμενε χώρε αρχίζουν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία η κατάσταση κάπως σχιζοειδής φαίνεται επειδή κάποιες φορές είναι ρασιτεχνική η προσέγγιση τους. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να καταλάβω ή αν υπήρξε απάντηση από τον κύριο Πίμπαλξ, αν θα γίνουμε πιο επιλεκτικοί στην επιλογή των κονδυλίων, στην απόδοση των κονδυλίων στο μέλλον. Και έπειτα από μια παρατήρηση τη κυρία Κέλλερ θέλω να λάβω αφορμή για την παρουσία του Ευρωκοινοβουλίου στο, στο Μπούζαν. Ε, στην Κινσάσα θυμάμαι, στην ε, κοινή συνάντηση με τις χώρε ΑΚΕ, είχαμε απαγορεύσει στον ε, κύριο Μισελ να εκπροσωπήσει τον, το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έτσι καλώς δεν εκπροσωπεί το. Και την αρμοδότητα αυτή την αποδώσαμε στον κυρία Άστον. Τώρα βλέπω η Πολωνική Προεδρία να αναλαμβάνει νέε αρμοδιότητε. Να απαγορεύει στο Ευρωκοινοβούλιο, α πούμε, να παρίσταται στι διαπραγματεύσει. Τι παράλληλε διαπραγματεύσει. Αυτό μα κάνει να θυμόμαστε το Μοτεσκέ που έλεγε ότι όποιο έχει στα χέρια του την εξουσία τήρει να την καταχράται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Είναι απολύτω απαράδεκτο, είναι γελίο. Είναι ντροπή, ντρέπεται κανεί να βλέπει το κοινοβούλιο να παρίσταται σε τέτοιου είδου συναντήσει. Θα πρέπει να ακούσουμε πολύ σοβαρού λόγου για να αποδεχτούμε κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν κάποια διευθέτηση του θέματο θα πρέπει να προβλεφθεί σε θεσμικό επίπεδο, ώστε να πάυσουν άπαξτε παντό αυτού του είδου συμπεριφορέ. Alors, euh, il existe un... Υπάρχει συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, και Κοινοβουλίου. Συμφωνία που ορίζει ξεκάθαρα ότι οι Ευρωβουλευτές έχουν ρόλο παρατηρητών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας απαγορεύσει κανείς την είσοδο ή την παρουσία μας. Νομίζω το πρόβλημα λοιπόν αυτό θα πρέπει σύντομα να λυθεί, γραπτός, και αν δεν αρκέσει αυτό, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς, θα το σημειώσουμε ίσως σήμερα και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να επιληθεί στην πράξη το θέμα. Μου έχει συμβεί και εμένα να μην μπορώ να μπω στη μια την άλλη αίθουσα. Το βρίσκω τελείως απαράδεκτο. Ε, δεν ξέρω λοιπόν τι μπορεί να γίνει πρακτικά. Ή αν το σημειώνει, εγώ το σκέφτομαι τώρα που το λέμε θα πρέπει να βρεθεί μια οριστική λύση στο θέμα αυτό. Κάθε φορά η κάθε προεδρία κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι απαράδεκτο. Απλώ διαπιστώνουμε το γεγονό μεν, αλλά αν είχαμε προηγουμένω λάβει τα μέτρα μα, ίσω να μην είχε διαθετηθεί το πρόβλημα εγκαίρω. Κύριε Γκέρεν, υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με το Συμβούλιο. Και το επαναλαμβάνω. Διότι ήδη είχα κάνει πρόταση να απευθύνουμε γραπτή επιστολή στο Συμβούλιο και να το καλέσουμε να αποσαφηνίσει κάποια ζητήματα. Όταν ε, συζητήσαμε το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων, το Συμβούλιο δεν εκπροσωπείται στι συζητήσει. Ενώ ω συνομοθέτη κάτι θα είχε να πει λογικά στην όλη διαπραγμάτευση. Ήταν δυσχερέστατε μάλιστα οι συζητήσει και δεν φτάσαμε και στο τέλο τη όλη προσπάθεια. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σαφή εμπειρία, ε, απουσία σχέσεων με το Συμβούλιο. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Εδώ θα πρέπει να υποτροπιάσουμε και να απευθύνουμε μια επιστολή στο Συμβούλιο, ώστε να βεβαιωθούμε ποιο ακριβώ κάνει τι. Και ώστε το Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται αξιοπρεπώς ή τουλάχιστον όπως δει στις διαπραγματεύσεις, διότι Νομίζω η αντίδραση έφυγε από τα όρια τη Επιτροπή μα. Θα έπρεπε ενδεχομένω ίσω το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε όλε τι διαπραγματεύσει διεθνού χαρακτήρα. Για τον επιπλέον λόγο ότι το Κοινοβούλιο βάσει τη Λισαβόνα έχει το δικαίωμα να πει την τελευταία λέξη για το όλο θέμα, τον τελευταίο λόγο. Μάλιστα, θα έρθουμε σε επαφή και με τι υπόλοιπε επιτροπέ, διότι όλε οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ έχουν το ίδιο πρόβλημα. Θα ετοιμάσουμε λοιπόν επιστολή τι ερχόμενε εβδομάδε και ίσω να θέσουμε και μία προθεσμία. Ιδάλω δεν θα γίνει. Αμένα μ' αρέσει να υπάρχει πλαίσιο χρονικό. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θέλουμε να ετοιμάσουμε μια επιστολή. Ίσως πρέπει να συζητηθεί στην διάσκεψη των Προέδρων. Στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα σας ενημερώσουμε. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Να βάλω και τα γυαλιά μου. Σημείο 18. Η σημερινή κρίση της ενέργειας έχει προβάλλει τι μεγάλε προσπάθειε που έχουν να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει τι ενεργειακέ τη ανάγκε. Με την αύξηση τη τιμή των ορεικτών καυσίμων, ένα αυξανόμενο αριθμό ε, γεωργικών πρωτονυλών γίνονται όλο και περισσότερο σπάνιε. Οπότε και πιο ακριβέ στην αγορά τη ενέργεια. Αυτή η αύξηση των πραγματικών τιμών κάποιε φορέ έχει σοβαρέ συνέπειε σε περιοχέ τη υπαίθρου και, του βιομηχανικού του κλάδου, αλλά και στην επιστημιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών. Για αυτό το λόγο, μια από τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ω προ τον προσανατολισμό τη αναπτυξιακή μα πολιτική αφορά την επεξεργασία και την υλοποίηση πολιτικών μέτρων, των οποίων ο στόχο θα είναι να εγγυηθούν την ε, εντυνόμενη χρήση της βιοενέργειας, ώστε να αντιμετωπίσουμε και την ένδια και την πείνα στον κόσμο. Παρουσιάζοντα αυτή τη μελέτη, η Επιτροπή μα θέλει να συμβάλλει στην όλη συζήτηση και να αποσαφηνίσει ποιε είναι οι πραγματικέ προκλήσει τη δύσκολη ισορροπία που επιδιώκουμε μεταξύ τη επίτευξη των στόχων από τη μια και τη ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη των φτωχών περιοχών του κόσμου. Έχουμε μαζί μα την ε, κυρία Στεφανή Βούντερ, ερευνήτρια ε, και συντονίστρια βιοενέργεια και γεωργία στο Οικολογικό Ινστιτούτο στο Βερολίνο, την οποία ευχαριστώ ε, που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας και στην οποία δίνει ευθύς αμέσως το λόγο. Το λόγο έχει η κυρία Βούντερ για ένα τέταρτο. Many thanks for that introduction. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή. Λέγομαι Στέφανη Βούντερ. Δεν είμαι από το Ινστιτούτο ΕΚΟ. Είναι διαφορετικό το Οικολογικό Ινστιτούτο στο Βερολίνο. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να παρουσιάσω τα κυριότερα ευρήματα σχετικά με τον αντίκτυπο της ε, πολιτικής βιοενέργειας της Ένωσης Αναπτυσσόμενης Χώρες. Πολλές έρευνες γίνονται σε αυτό το τομέα, κυρίως για τα βιοκαύσιμα. Εγώ ε, ε, ήρθα από, έρχομαι από την Επιτροπή Ένβη, που εξετάσαμε εκεί τα θέματα των βιοκαυσίμων Τώρα θα μιλήσουμε πιο πολύ για την ξυλώδη βιομάζα. Οπότε αυτό που θα παρουσιάσω τα επόμενα 15 λεπτά ε, θα κοιτάξω να συντομεύσω για να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Θα παρουσιάσω τη βάση της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα βιοενέργειας, να δούμε την ε, ζήτηση σε ξυλώδη βιοενέργεια, μετά να δούμε τις ροές του εμπορίου και το ρόλο των αναπτυσσομένων και το βασικό αντίκτυπο των στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες σε ό,τι αφορά ασφάλεια, τοπική ενεργειακή ασφάλεια, πρόσβαση στο, στη γη και στο νερό, περιβαλλοντικός αντίκτυπος και συμπεράσματα. Όπως ξέρετε, η οδηγία ανανεώσιμων, του, ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του 2009 ήταν η βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της βιοενέργειας στην Ένωση που εξακολουθούμε να παραβλέπουμε σήμερα. Χωρίζεται σε 20% ανανεώσιμους στόχους, ε, ε, ε, πηγές ανανεώσιμες το 2020 και 10% καύσιμα για τις μεταφορές από ανανεώσιμες πάλι μέχρι το 2020. Στόχος βιοκαυσίμων δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον αυξανόμενο για την ξυλώδη βιομάζα, αξιοσημείωτο. Χρησιμοποιείται η βιομάζα αυτή ξυλώδης κυρίως ε, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ε, ψήξη, θέρμανση. Ε, έχουμε βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, τώρα βιοκαύσιμα από ξυλώδη βιομάζα. Αυτά είναι η δεύτερη γενιά και τότε και τα βιοκαύσιμα θα είναι μια εναλλακτική, αλλά σε μικρή κλίμακα για την χρήση ξυλόδους βιομάζας. Τώρα, περνώντας στο, σε εθνικά προγράμματα δράσης που υπέβαλαν όλα τα κράτη, εδώ η ζήτηση και οι πολιτικοί στόχοι στα κράτη-μέλη δεν μπορούν να καλυφθούν από την εγχώρια παραγωγή στην Ένωση, αλλά θα καλυφθούν από εισαγωγές από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι δύσκολο να δούμε σε ποιο βαθμό θα, δώσουν, θα παίξουν ρόλο οι φοιτίες, οι εκτάσεις. Πάντως θα είναι ο ρόλος τους πολύ σημαντικός. Μιλάμε για ζήτηση. Οι εισαγωγέ τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από πού θα προέρχονται, αυτή είναι μια ερώτηση. Και είναι ενδιαφέρον γράφημα αν δούμε τις πράσινες περιοχές όπου υπάρχει αυξανόμενο δυναμικό συγκομιδής κυρίως Νότια Αμερική, Ανατολική Ευρώπη και Αφρική και μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας. Για την Ευρώπη βλέπουμε σταθεροποιημένη τη συγκομιδή, αλλά υψηλή ζήτηση ακόμα εξακολουθεί να είναι υψηλή. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εισαγωγή βιομάζας. Άλλο γράφημα εδώ που δείχνει κάποια παραδείγματα μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, έργα. Παραδείγματα βλέπουμε Γκάνα, Κονγκό, Μοζαμβίκη. Αυτά είναι έργα μεγάλης κλίμακας και από εκεί μπορεί να προέλθει ξυλώδης βιομάζα. Αναλύσαμε τον αντίκτυπο. Όταν μιλούμε για αντίκτυπο είχαμε υπόψη μας ε, δυνητικά ωφέλη και ανησυχίες προβλήματα Φαντάζεστε κι εσείς ότι είναι δύσκολο να εντοπίσουμε το συγκεκριμένο αντίκτυπο της πολιτικής ένωσης για την βιοενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και διότι είναι πολύ μεγάλη γενικότερα η ζήτηση στην αγορά, όχι μόνο στην ε, αγορά της Ένωσης, αλλά και επειδή υπάρχουν άλλες χρήσεις για τα έπιπλα, παραγωγή χάρτου, όπου χρησιμοποιείται ξυλώδης βιομάζα και σε άλλους τομείς και αυτά δρούν ανταγωνιστικά στην ίδια, μέσα στην ίδια αγορά. Θα σας δείξω λοιπόν κάποια γενικότερα στοιχεία εις ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που εξετάζουμε και μετά όπου είναι δυνατόν θα καταδείξω κάπως καλύτερα το ζήτημα μέσα από παραδείγματα, κυρίως από την Αφρική, γιατί αυτή είναι η περιοχή που εξετάζουμε ως επιτοπλίστων. Ο πρώτος τομέας αντικτύπων ήταν η πρόσβαση στη γη των ε, αγροτικών κοινοτήτων στις ΓΕΕΣ. Όπως στις συζητήσεις που κάναμε ε, για τον τομέα των βιοκαυσίμων, υπάρχει ο φόβος της καταπάτησης γεών, υδάτων, μεγάλης κλίμακας, ε, έργα από εξωτερικούς επενδυτές και το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι συμφωνίες ε, καταλαμβάνουν και δημόσιες γέες, ε, κοινοτικές και αυτές οι κοινότητες συνήθως δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας ε, επίσημους. Μιλάμε για την Αφρική, 2 με, όπου 2 με 10% των γεών στην Αφρική μόνο ε, έχουν επίσημους τίτλους. Οπότε καταλαβαίνετε την έκταση του προβλήματος. Και επίσης ε, η διαβουλεύση με τις κοινότητες συχνά είναι ανεπαρκείς ε, ή δεν υπάρχει αρκετή, αρκετά ικανοποιητική εκπροσώπηση. στο Καμερούν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν κάνει συζητήσεις με την κοινότητα όταν παραχωρούν γη στους επενδυτές. Το πρόβλημα με την επίσημη αξίωση και τους τίτλους είναι ότι οι κοινότητες συχνά αποκλείονται από τα ωφέλη που προκύπτουν. Ε, θα μπορούσαμε εδώ να μιλήσουμε για την απασχόληση, όπου ναι μεν δημιουργούνται κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά αυτοί που επηρεάζονται αρνητικά ε, δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι με αυτούς που κράτησαν τη δουλειά. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ιδιαίτερα στις φοιτίες οι εξοπλισμοί και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται απαιτούν λιγότερο προσωπικό για να τα χειρίζεται τα μηχανήματα. Στη Μοζαμβίκη βλέπουμε ότι Ήταν παροδική η απασχόληση ε, και χρειάστηκαν νέες διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να αποκομίσουν κάποια ωφέλη από τις επενδύσεις στον τομέα των σχολείων, πρόσβαση, έργα για πρόσβαση στο νερό κλπ. Η πρόσβαση στο νερό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Προφανώς ένα βασικό ζήτημα είναι ότι συνήθως απαιτούν οι φοιτίες μεγάλες ποσότητες νερού στο ε, ρευκάλιτο, για παράδειγμα. Επίσης τα ζυζανιοκτώνα ε, που χρησιμοποιούνται, οι εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται ε, όταν ετοιμάζεται η φυτεία και γίνεται η εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσουν σε ρήπανση των τοπικών υδάτινων πόρων. Επίσης τα δικαιώματα στο, στα ύδατα όπως και στις γέες δεν είναι επίσημα και υπάρχουν πρόβλημα και μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Η ασφάλεια, η επισητιστική ασφάλεια είναι σημαντικό θέμα. Οι χώρες που επηρεάζονται από την επισητιστική ασφάλεια είναι οι δυνητικά εξαγωγικές χώρες. Ο άμεσος ανταγωνισμός μεταξύ φυτιών βιομάζας και ε, γόνιμων γεών ε, είναι ένα αίτιο του προβλήματος. Πολλές φορές υποβαθμισμένες γέες μπορεί να αποτελούν μια λύση ανηφιτίες για την παραγωγή ξυλόδους βιομάζας είναι σε μη γόνιμες γέες, είναι μικρότερο το πρόβλημα. Αλλά είδαμε ότι δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν ποτέ αυτές οι υποβαθμισμένες γέες, γιατί εκεί το κόστος είναι υψηλότερο και η απόδοση μικρότερη. Οπότε συχνά δεν χρησιμοποιούνται. Ε, η αύξηση στις τιμές των τροφίμων ε, είναι επίσης ε, μια απόρρεια των, ε, της παραγωγής βιοκαυσίμων και αν χρησιμοποιηθούν οι περιοχές αυτές για άλλες χρήσεις, συνήθως είναι βιο ε, λογικά τρόφιμα. Επίσης, ε, με την παραγωγή ξυλόδους βιομάζας χρησιμοποιείται για κάποιες δεκαετίες η γη, δεν μπορεί δηλαδή να αλλάξει γρήγορα και να πάμε στα ε, βιοκάψιμα. Επίσης έχουμε με αυτόν τον τρόπο πόλια εισοδηματικών ευκαιριών. Ε, τώρα, η, σε, τοπικό επίπεδο η ενεργειακή ασφάλεια. Συνήθως έχουμε υψηλή εξάρτηση ε, σε, από πηγές ενέργειας με βάση το ξύλο. Στην Αφρική είναι 89%, στην Ασία 81% και στη Λατινική Αμερική 66% η εξάρτηση από ε, ενεργειακές πηγές με βάση το ξύλο. Υπάρχει λοιπόν μια σύγκρουση εδώ στους στόχους ε, αν οι χώροι παραγωγής ε, ε, παρεκτοπίσει την χρήση ενεργειακών πόρων με βάση το ξύλο που πλέον δεν θα καλύπτουν τον τοπικό πληθυσμό. Τέλος, περιβαλλοντικός αντίκτυπος ε, είναι πολύ μεγάλη γκάμα εδώ. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο όπως η ένταση της παραγωγής, η κλίμακα, ε, τα είδη των δέντρων που θα χρησιμοποιηθούν, συστήματα συγκομιδής και πολλοί άλλοι παράγοντες. Αλλά βέβαια μπορεί να υπάρξουν και ωφέλη, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την παραγωγή βιοκαυσίμων, με ετήσια, μονοετήφητα, ε, για την παραγωγή βιοκαυσίμων, γιατί η δάσωση επηρεάζει, μπορεί να μειωθούν επίσης οι δασικές πυρκαγιές ή ο κίνδυνος για αυτές, μπορεί να μειωθεί η απορροή υδάτων και η απώλεια ε, Ζημάτων. Υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις όμως ε, από ψήλωση, υποβάθμιση των δασών, άμεση-έμεση μετατροπή γεών, που μετατρέπεται σε φυτίες και φυτίες σημαίνουν χαμηλότερη βιοπικιλότητα και αξία των γεών και καλλιεργών και, καλλιεργιών και πολλά άλλα αρνητικά. Για τα συμπεράσματα, αυτό που είναι ενδιαφέρον και έχει άμεση σχέση με την αποψήλωση είναι ε, το πολιτικό πλαίσιο ο ορισμός ε, του ΦΑΟ των δασών είναι τέτοιος, ώστε εν μέρει και τις φυτίες. Να διαβάσω τον ορισμό. Τα δάση σύμφωνα με τον ΦΑΟ είναι γες που καλύπτουν περισσότερο από μισό εκτάριο με ε, πάνω από 5 μέτρα ψηλά δέντρα και ε, το φύλλωμα, το θόλο του δέντρου με συγκεκριμένες διαστάσεις. Αυτό που γίνεται, που ε, συμβαίνει με τον ορισμό, είναι ότι η αποψήλωση δεν ε, συνυπολογίζεται. Γιατί κόβουμε τα δάση, φτιάχνουμε φυτεία και εξακολουθεί να είναι δασική η περιοχή σύμφωνα με τον ορισμό. Και το πρόβλημα είναι ότι ο ορισμός του ΦΑΟ χρησιμοποιείται μετά στο UNFCCC, δηλαδή στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και την πολιτική για το κλίμα. Και έτσι διευρύνεται η περιοχή που καλύπτεται από δάση. Επίσης ε, υπάρχουν ασθενείς μέσα ε, διακυβέρνησης ε, για τα δάση. Μόνο το 18% έχει πιστοποιηθεί, μόνο για το 18% γίνεται πιστοποιημένα καλή διαχείριση. Και δεν υπάρχουν δεσμευτικά, δεσμευτικές προϋποθέσεις για την αηφορία, για την χρήση ε, στέρεας και αέριας βιομάζας. Ε, τώρα, για τα συμπεράσματα βλέπουμε ότι προφανώς είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε συγκεκριμένο αντίκτυπο της πολιτικής της Ένωσης για τη βιοενέργεια, αλλά πέρα από τον αντίκτυπο σε επίπεδο έργου και οι επιπτώσεις ως επιτοπλίστων έμεσες αλλά είναι πολύ σοβαρές και με την αυξημένη ζήτηση έχουμε αύξηση της τιμής του ξύλου και έτσι έχουμε αυξημένη πίεση στα οικοσυστήματα και τα ε, οικοσυστήματα και ε, συγκρούσεις στη χρήση της γης και επηρεάζονται έτσι και οι τιμές των τροφίμων. Αυτό πάλι επηρεάζει ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι αυτά τα έργα είναι μακροπρόθεσμα, μακράς διάρκειας και μπορεί ενδεχομένως να ε, βλάψουν την πρόσβαση στη γη και στο νερό και στην ενέργεια και την ασφάλεια τροφίμων μπορεί να την επηρεάσουν για δεκαετίες αρνητικά και υπάρχει και πρόβλημα διακυβέρνησης. Αυτά λοιπόν που θα ήθελα να συνοψίσω είναι οι τρεις ανάγκες αν θέλετε και πάνω εκεί να συζητήσουμε οι τρεις προσεγγίσεις για να δούμε την αρνητική, το πρόβλημα του αρνητικού αντίκτυπου. Πρώτον, χρειάζεται να μειωθεί το οικολογικό αποτύπωμα της Ένωσης προς μεγαλύτερη αποδοτικότητα ενεργειακή και αποδοτικότητα πόρων, γιατί έχουμε μεγαλύτερο αποτύπωμα από τη διαθέσιμη έκταση, αν θέλετε, την επικράτεια της Ένωσης. Αυτό πρέπει να είναι ένας στόχος. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό οι αναπτυσσόμενες χώρες να υποστηριχθούν για να δημιουργήσουν μηχανισμούς καλής διακυβέρνησης και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ε, στη γη, ε, διακυβέρνηση, ε, διαχείριση δασικών πόρων κλπ. δασών και να διευρύνουμε τη συζήτηση για τα πρότυπα βιωσιμότητας και αηφορίας πέρα από τα περιβαλλοντικά για να συμπεριλάβουμε επισκεπτική ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια, πρόσβαση στις, ε, στη γη, να συμπεριλάβουμε τη βιομάζα και όχι μόνο τα βιοκαύσιμα για τη μεταφορά, τις μεταφορές, στα πρότυπα της αηφορίας, όπως το συζητάμε, αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Και επίσης ε, θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουν όποιες αλλαγές ε, στην, έμεση χρήση της γης, να συμπεριλάβουν και τη βιομάζα και όχι μόνο τα βιοκαύσιμα και εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ την κυρία Βούντερ και ζητώ και συγγνώμη γιατί έχω την εντύπωση ότι ε, έφυγαν οι συνάδελφοι γιατί είχαν άλλες δουλειές προφανώς να κάνουν. Εσείς όμως ε, θίξατε ένα απίστευτα σημαντικό θέμα, σημαντικό όχι μόνο για τους πολιτικούς στον τομέα της ανάπτυξης, αλλά για όσους ε, ασχολούνται με μέσο και μακροπρόθεσμες πολιτικές. Και καλό θα ήταν να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό για να τα ακούσουν περισσότεροι γιατί είναι σημαντικό. Όπως είπαμε, μακροπρόθεσμα δεν ε, έχει να κάνει μόνο με το επίπεδο και την πολυτέλεια μιας ζωής μας, αλλά, της ζωής μας, αλλά για την ποιότητα των τροφίμων και πολλά άλλα σημαντικά. Ευχαριστώ. Ναι, και λυπάμαι, λυπάμαι ιδιαίτερα για την απουσία αυτή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Λυπάμαι που η αίθουσα είναι άδεια. Βρίσκω πως ε, δεν δείχνει αρκετό σεβασμό προς το πρόσωπό σας. Και βέβαια για το κατά πόσο ενδιαφέρονται οι βουλευτές ε, για το θέμα σας. Ε, αν δεν τους ενδιαφέρει το θέμα θα μπορούσαν να έχουν επιλέξει άλλη επιτροπή. Είναι το μόνο που μπορώ να πω. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Λαμπέρ από τη Σχετική Γενική Διεύθυνση και μετά θα κλείσουμε τη συνεδρίαση και θα στείλουμε ένα μήνυμα σε όλα τα μέλη αυτής της ε, Επιτροπής, γιατί πραγματικά είναι ντροπή να είμαστε τόσο λίγοι. Κύριε Λαμπέρ, έχετε το λόγο. Είμαι από την ε, Γενική Διεύθυνση ε, Ανάπτυξης και πρέπει να πω πως βρήκα την ε, εκθέση σας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είναι ένα θέμα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική μας Διεύθυνση ε, δίνει ιδιαίτερη σημασία. Θα συμμεριστούμε απόλυτα την ανάλυση κινδύνου που έχετε κάνει και τα όσα είπατε. Ξέρουμε ποιος είναι ο θετικός αντίκτυπος και ποιος ο αρνητικός, όχι μόνο για τα περιβαλλοντολογικά θέματα, για την αποψήλωση, για την καταστροφή της βιοπικιλότητας, που είναι μεγάλες απώλειες, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο και οικονομικό βέβαια. Γιατί είναι γη που δεν έχει πρόσβαση στην, σε νερό, που δεν εξασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό. Νομίζω ότι θα πρέπει να παραπέμψουμε άμεσα στο τι έχουμε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ. Εμείς λάβαμε υπόψη τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα επόμενα project που έχουμε για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα και θα τα λάβουμε δεόντως υπόψη. Κάνουμε κάποιες προσπάθειες και σε νομοθετικό επίπεδο, στις ευρωπαϊκές ε, ρυθμίσεις έτσι ώστε η αεριώδης και η στερεά ε, βιομάζα να εξεταστεί όπως πρέπει και βέβαια εξετάζουμε τι γίνεται από, τους, από τις χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του αγαθού. Τώρα, ποιε είναι οι απαντήσεις που θα έπρεπε να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Καλύτερη διακυβέρνηση και σε τοπικό επίπεδο. Μια αμυντική στάση, η οποία θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε όλα αυτά τα αγαθά και τους πόρους γιατί υπάρχει και το αναπτυξιακό πρόβλημα που έχει δείξει πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για την διαχείριση των δασών, κάποια στοιχεία θα πρέπει να αναφέρουμε, αξίζει τον κόπο. Έχουμε τον RED το μηχανισμό RED που είναι η μείωση των εκπομπών άνθρακα που προκύπτει από την αποψήλωση των δασών, στα πλαίσια των προσπαθούν που κάνουμε για την αλλαγή του κλίματος γιατί τα αέρα του θερμοκηπίου όντως συνδέονται με την εξαφάνιση των δασών στον πλανήτη και για τις ενδιαφερόμενες χώρες ε, η προσπάθεια γίνεται να δουν για ποιο λόγο χάνονται τα δόση. Κακή διαχείριση, ε, έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης, έλλειψη προσπάθειας δάσωσης ο ορισμός από τον ΦΑΟ του τι είναι δάσος εμπίπτει στον κλάδο αυτό. Εμείς έχουμε και τον μηχανισμό RED που μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη και το παγκόσμιο, ε, την Παγκόσμια Τράπεζα προσπαθεί να βελτιώσει την διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου. Έχουμε λοιπόν και το Forest Law on Governance and Trade, το νόμο FLECT ε, για την διαχείριση των δασών και την εμπορία των δασικών προϊόντων για την νόμιμη εξαγωγή ε, δασικών προϊόντων, έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και να λαμβάνουμε υπόψη και την κοινωνικο-οικονομική πτυχή αυτής της εμπορίας η πρωτοβουλία φλέκτη e είναι 100% ε, ευρωπαϊκή. Η Λιβερία αναφέρεται στο έργο αυτό γιατί παράγει βιομάζα που την εξάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία από τις χώρες που υπέγραψαν μία ε, συνθήκη ΦΛΕΚΤ. E Βρίσκεται στην φάση της επικύρωσης υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή το θέμα στα πλαίσια της ανεπτυξιακής της πολιτικής έτσι ώστε κάποια θέματα να αποσυμφορηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βούντερ, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση αυτή. Δεν άκουσα ερώτηση για το θέμα αυτό, αλλά ενδεχομένως το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες point, uh, more detailed look what, what else Ίσως περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα γίνει. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στο FLECT. Είναι μια καλή ευκαιρία για τη διαχείριση και τη λέξη αυτή που είναι τόσο της μόδας, να σας πω πως όσο πιο πολύ ε, λεπτομερώς περιγράφεται, τόσο περισσότερα αποτελέσματα φέρνει, τόσο πιο πολύ είναι αυτοί που ευνοούνται από τη χρήση της. Μιλάμε λοιπόν για ε, ανεφοδιασμό, για τα κτλ. Αλλά σας ευχαριστώ για ε, το σχόλιο, το σχετικό. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων. Ο κύριος Παγίου βρίσκεται στη θέση του. Όχι. Είμαστε στο 19. Ο κύριος Βάγκλη έχει σειρά για να πάρει το λόγο. Α, μάλιστα, πρόκειται για σφάλμα. Η κυρία Μανσίτη φτάνει. Όπου να είναι φτάνει. Δύο λεπτάκια και θα είναι εδώ. Και για να κλείσουμε, έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, στην ε, ανταλλαγή απόψεων για τον δομημένο, διαστρωμένο διάλογο με τους μη κρατικού παίκτες και με τις τοπικές αρχές, έτσι ώστε να συζητήσουμε τις βασικές μας συστάσεις. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν έχει ε, ετοιμάσει ένα έργο εργασίας με συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον αυτού του διαλόγου και τα συζητήσαμε 9 και 10 Νοεμβρίου στα πλαίσια του διαλόγου αυτού. Δεν ξέρω εάν έχουμε βουλευτή στην αίθουσα. Δύο βουλευτές βρίσκονται εδώ. Μα ειλικρινά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Euh, Θέλετε να ζητήσω να αναβληθεί. Euh, euh- Κυρία Σνίβερ, τι επιθυμείτε εσείς. Frau Schnieber, bitte. Äh, äh, τι περιμένετε από εμάς να περιμένουμε να φτάσει το συγκεκριμένο άτομο ή να το αναβάλουμε. Να κλείσουμε. Κλείνουμε. Λοιπόν, είναι λίγο αποθαρρυντικό. Θα σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ όλους. Θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε. Αλλά βεβαίως δεν είναι ευχάριστο για κανέναν. Κλείνω λοιπόν τη συνειδίαση νωρίτερα από το ε, προβλεπόμενο και σας εύχομαι καλό βράδυ.